So, ladies and gentlemen, distinguished experts. Κυρίε και κύριοι, διακεκριμένοι εμπειρογνώμονε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμμετέχοντε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να σα καλωσορίσω στη δημόσια αυτή ακρόαση για την επίπτωση που έχουν ε, οι ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές και στη συνέχεια θα τους αποκαλούμε ενδοκρινικούς διαταράκτες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσια Υγεία, Ασφάλεια Τροφίμων και Επιτροπή Αναφορών Συνδερμανών, την ακρόαση αυτή. Θα ξεκινήσω με κάποιες πρακτικές πληροφορίες. Προβλέπετε και παρέχετε διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Επιτροπής μας. Πλην νεοστονικών και Σλοβενικών. Δηλαδή, Εστονοί και Σλοβενοί συνάδελφοι, λυπούμε, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα, θα πρέπει να μιλήσετε άλλη γλώσσα. Τα μέλη του πάνελ θα έχουν ο καθένας στη διάθεσή του 10 λεπτά και μετά από κάθε πάνελ θα έχουμε ανταλλαγή ε, απόψεων, συζήτηση με τους παρισταμένους. Επίσης, η ακρόαση αυτή μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Το θέμα της σημερινή ε, δημόσιας ακρόασης είναι οι ανησυχίες που αφορούν την ασφάλεια των χημικών ουσιών που αποκαλούμε ενδοκρινικούς διαταράκτες. Έχουν ε, γίνει δεκτές εδώ στην Επιτροπή μας πολλές αναφορές για το θέμα αυτό που δείχνουν πόσο έντονες είναι ανησυχίες μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Δύο θα είναι τα πάνελ της ακρόασης. Το πρώτο θα δει κατά πόσον η προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ρύθμιση των εθνικών μεταλλακτών είναι η ενδεδειγμένη και αν χρειάζονται αλλαγέ στο μέλλον. Και το δεύτερο θα αξιολογήσει την κατάσταση τη επιστημονική γνώση για τα αποτελέσματα ε, τη τι επιπτώσει των ενδοκρινικών διαταρακτών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Ευχαριστώ και εύχομαι μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Πρώτο πάνελ. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίζει ε, τα πράγματα με το σωστό τρόπο. Έχουμε τρεις εμπειρονόμους, τον κύριο Κόνορ Κλέναγκαν, καλώς ήρθατε, την κυρία Άλις Μπέρνερ, καλώς ήρθατε, και την κυρία Πασατσιγκότη. Χαίρομαι που ήρθατε εδώ. Σας καλωσορίζω και τους τρεις. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κλέναγκαν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ε, ευχαριστώ για την πρόσκληση στη σημερινή ακρόαση. Θα ήθελα να σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση του οργανισμού για τα χημικά, σε ό,τι αφορά τους διαταράκτες. Να σας εξηγήσω καταρχάς λοιπόν τι κάνει ο ΕΚΑ, ο Οργανισμός Χημικών. Εφαρμόζει τον κανονισμό REACH, το CLP, τον κανονισμό για τα βιοκτώνα και την εκ των προτέρων, ε, ε μάλλον τη συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωση, το prior informed consent. Συνεργαζόμαστε με τα κρατημέλη, την Κομισιόν και τους διαφόρους άλλους ε, ενδιαφερόμενους. Για την εφαρμογή αυτών των ε, νομοθετημάτων συλλέξαμε πάρα πολλές πληροφορίες, μοναδικός ο πλήθος των πληροφοριών για τα χημικά και οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να, να αξιολογήσουμε τους κινδύνους των χημικών ουσιών και να εφαρμόσουμε μέτρα ασφαλείας, προστασίας. Είτε ρυθμιστικά μέτρα ελέγχου ε, που γίνονται οι έλεγχοι αυτοί από, τους αρχές, από τις αρχές ή με βάση τους κινδύνους των χημικών ελέγχους και μέτρα ασφαλείας από τις ε, επιχειρήσεις. Και βλέπετε ότι έχουμε και πολλές νέες, ε, πολλές νέες τομείς εργασίας Δηλαδή επεκτείνεται ε, το πεδίο, το πεδίο που μας απασχολεί και ο ρόλος μας. Ποιες είναι βασιλικές διαδικασίες ή καταχώρηση, πληροφορίες ε, δίνονται από τον ΕΚΑ, συλλέγουν οι ε, κλάδοι της μηχανές πληροφορίες και εξασφαλίζουμε τη διαχείριση των κινδύνων. Υπάρχει αξιολόγηση και έπειτα υπάρχει και η διαχείριση των κινδύνων, η αδειοδότηση, οι περιορισμοί. Βασικά πρόκειται για μέτρα διαχείρισης κινδύνων. Πώς λοιπόν ρυθμίζονται οι ενοκρινικοί διαταράκτες. Ο ΕΚΑ εφαρμόζει αυτή τη στιγμή μια ολοκληρωμένη ρυθμιστική στρατηγική για τη διαχείριση όλων των ουσιών που έχουν καταχωριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπα και πριν ότι έχουμε μια τεράστια βάση δεδομένων. Στην περίπτωση των ενδοκρινικών διαταρακτών μελετάμε ε, τις ουσίες που μπορεί να εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Βλέπουμε ποιες είναι οι επικίνδυνες ιδιότητες, χρήση, έκθεση των νοσιών για να δούμε ποιες είναι οι ουσίες προτεραιότητας για τις οποίες χρειάζεται να ληφθεί δράση αυτή είναι η διαδικασία του screening. Τα δεδομένα της καταχώρησης και άλλες πληροφορίες μας βοηθούν να εντοπίσουμε δυνητικούς ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες. Μελετούμε τα στοιχεία και εντοπίζουμε υποψήφιες ουσίες που θα πρέπει να μας απασχολήσουν περαιτέρω. Εστιάζουμε επίσης ε, στις ε, πιο σημαντικές από αυτές τις ουσίες. Έπειτα, παραγωγή περαιτέρω πληροφοριών και αξιολόγηση. Η διαδικασία αξιολόγηση μας βοηθά να συλλέξουμε πρόσθετες πληροφορίες για κάποιε ουσίες. Όταν ε, δεν αρκούν οι πληροφορίες καταχώρησης, ε, υπάρχει και ένα σχέδιο δράσης ε, για την αξιολόγηση. Και σε αυτό το σχέδιο δράσης έχουμε 82 ουσίες δεν είναι εύκολο να σε μία αξιολόγηση. Υπάρχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που τρέχει τα κράτη-μέλη. Και όταν ε, παράγονται περισσότερες πληροφορίες, η βιομηχανία υποχρεωμένη να τις ε, λάβει υπόψη. Υπάρχουν συζητήσεις ε, σε σχέση με τον ορισμό ενδοκρινικού διαταράκτη. Έχει η Παγκόσμια Οργάνωση υγείας ε, την, ε, τον ορισμό λέξογενείς ουσίες που επηρεάζουν, αλλοιώνουν τις λειτουργίες του κλινικού συστήματος και ε, δημιουργούν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία ενός οργανισμού υποπληθυσμών αυτού. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη το έργο του ΟΣΑ και υπάρχει και μια ομάδα στο πλαίσιο του Κοινού των Ερευνών και της ΕΦΣΑ που γνωμοδοτούν. όλοι αυτοί μας βοηθούν να δούμε τι περαιτέρω πληροφορίες χρειάζονται για να καταλήξουν στο κατά πόσο μια ουσία είναι ή δεν είναι ενδοκρινικός διαταράκτη. 80% των συζητήσεων αυτό αφορά και μας βοηθάει πάρα πολύ και η δουλειά που κάνει ο ΣΑ, είπα. Σε ό,τι αφορά το REACH για την ε, διαχείριση κινδύνων. Θέλουμε να προωθήσουμε την υποκατάσταση και να ε, εξασφαλίσουμε υψηλά επίπεδα προστασίας μέχρι να βρούμε μια εναλλακτική ουσία. Έχουμε συμπεριλάβει 12 ουσίες ε, στον κατάλογο ε, υποψηφίων να έχουν τέτοιες διατερότητες, φαινόλες και φθαλάτες. Οι ουσίες που έχουν ε, ιδιότητε διατάρξης του δοκνικού συστήματο του συστήματος ήδη υπόκειται σε περιορισμού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του REACH ε, για ως βάση για την ανάπτυξη δράση στο πλαίσιο και άλλων νομοθετημάτων και υπάρχουν διάφορα νομοθετήματα σχετικά και έτσι έρχομαι ε, στα βιοκτώνα και στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τους σχετικούς κανονισμούς. Τα κριτήρια ενδοκρινικής διαταραχής για τα βιοκτώνα μελετούνται, ισχύουν για τα βιοκτώνα και μελετούνται για ε, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Βασίζονται στις οδηγίες ε, του, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, δηλαδή η ίδια βάση που χρησιμοποίησαμε για την ε, για τον εντοπισμό και αυτοποίηση ενδοκρινικών διατακτών. Και μαζί με την ΕΦΣΑ και το Κέντρο Ερευνών αναπτύσσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την ε, ε, εντοπισμό ε, τέτοιων ενδοκρινικών διατακτών βάσει κινδύνων. Έχουμε σε επαφή και έχουμε διαβουλεύσει με τους ενδιαφερομένους φορείς ό,τι αφορά ε, την, ε, τα κριτήρια αυτά. Είναι μια δημόσια διαβούλευση και τον Ιούνιο του 2018 θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα για να ολοκληρώσω. Το REACH δίνει πληροφορίε, δίνει εργαλεία για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση ενδοκρινικών διαταρακτών, αλλά υπάρχει δυνατότητα βελτίωση σε ό,τι αφορά την ποιότητα και ποσότητα των δεδομένων και των καταχωρήσεων και εξετάζουμε ε, τρόπους για να επιταχύνουμε τη διαδικασία ταυτοποίησης ε, που μπορεί να είναι ιδιαίτερα μακρά, μακροχρόνια γιατί πολλές φορές πρέπει να ζητήσουμε ε, πληροφορίες επιστευτικές και αυτό απαιτεί κάποια διαδικασία και κάποιο χρόνο. Επίση, η βιομηχανία πρέπει να εξασφαλίσει την ασφαλή χρήση και να στηρίξει την υποκατάσταση της ουσία. και οι αρχές έχουν επίσης τη δυνατότητα να εισαγάγουν μέτρα διαχείρισης κινδύνων ε, και το ΕΚΑ έχει ήδη στο πλαίσιο του ΡΙΤΣ ε, εντοπίσει και επιβάλλει περιορισμού σε πολλές ουσίε που χαρακτηρίζονται κοινωνική διατάξη. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε. Ερωτήσεις και παρατηρήσεις στο τέλος ε, του πάνελ. Οπότε τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπέρναν, ε, στην κυρία συγγνώμη ε, για την παρουσίασή της. Σας ευχαριστώ. Μόλις ακούσαμε λοιπόν από έναν ρυθμιστή, την ΕΚΑ, και εγώ θα σας μιλήσω από την νομική οπτική και μου ζητήθηκε να παρουσιάσω πώς η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ρυθμίζει τους διαταραχτές, όχι μόνο με το ΡΙΤΣ, Κάπως ε, βέβαια δύσκολο σε 10 λεπτά να το κάνω αυτό. Ε, βεβαίως ε, θα είναι μια επισκόπηση. Um, just a, a few words on, on Claritas, the organization I, I work for. Um, η Client Earth είναι ο οργανισμός για τον οποίο εργάζομαι. Όπως γνωρίζετε δεν μπορούμε πάντοτε να προσλάβουμε έναν νομικό, ενώ η χημική βιομηχανία μπορεί κάλλιστα να το κάνει αυτό. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ρυθμίσει ε, το θέμα. Πρόκειται για θέμα υγείας και περιβάλλοντος. Επειδή οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμα καταλήξει, να σας πω τι έχουμε εδώ. Έχουμε χημικές ουσίες που μπορεί να περιορίσουν, να αναστείλουν το ενδοκρινικό το σύστημα, το δικό μας ή των ζώων, με διάφορες ε, και πολλές ε, επιρροές και παρενέργειες. Άρα λοιπόν στα θέματα υγείας και περιβάλλοντος η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ε, κάνει προληπτικές ενέργειες μέσα στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος ε, πλαισίου για το περιβάλλον. Ε, απόφαση που ελήφθη από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο περιλαμβάνεται εκεί μια ολόκληρη μεγάλη παράγραφος για το πώς πρέπει να περιοριστεί η έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες. Το 2016 το Συμβούλιο θύμισε στην Ένωση αυτή της, την υποχρέωση. Πρώτα όμως να σα πούμε πώς ε, λειτουργούν αυτά τα χημικά. Έχουμε πρώτον την ε, διαπίστωση του προβλήματος που είναι βασικά ε, ζήτημα ποιες είναι οι ιδιότητες ενό ε, χημικού οι οποίες δεν αλλάζουν ανάλογα με την ε, ε, τη χρήση και το δεύτερο ζήτημα, το δεύτερο βήμα είναι η διαχείριση του προβλήματος. Δηλαδή, τι απόφαση θα λάβει το Συμβούλιο από αυτού, αν δηλαδή θα ρισκάρει ή όχι Θέλουμε να έχουμε το παράδειγμα των καρκινογόνων ουσιών. Γενικά, πώς αυτές ρυθμίζονται στο, ε, στην Ένωση. Πρώτα έχουμε το βήμα του, της ταυτοποίησης. Ε, αυτό γίνεται με έναν κανονισμό αυτόν της ταξινόμησης ε, και το Συμβούλιο έτσι αποφασίζει ότι το τάδε ας η τάδε χημική ουσία πρέπει να ταξινομηθεί στις καρκινογόνες και αυτή είναι η πρώτη και κεντρική οδηγία που εναρμονίζει ε, το είδος των χημικών. Ξεκινάμε από τα δεξιά, μετά από την πρώτη ταξινόμηση. Έχουμε πρώτη την οδηγία περί παιχνιδιών, όπου απαγορεύεται η χρήση τους, παρομοίως για τα καλλιτικά, παρομοίως για τους, τις ιατρικές συσκευές. Ε, δεν είναι το τέλειο σύστημα για τις καρκινογόνες ουσίες, ε, θα πρέπει να εξετάσουμε την εφαρμογή όλων αυτών. Υπάρχουν πολλές ε, εξαιρέσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ε, γενικό σύστημα. Πώς δουλεύουμε λοιπόν για τους ενδοκρινικούς ε, διαταράκτες. Όπως βλέπετε, στον ε, στάδιο του εντοπισμού τους και της αναγνώρισής τους δεν έχουμε μια συγκεκριμένη ταξινόμηση. Στην πρώτη οδηγία ταξινόμησης ε, ε, σήμανσης και συσκευασίας, όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, υπάρχει το REACH που επιτρέπει τον εντοπισμό και την αναγνώριση των ενδοκρινικών διαταρακτών ως ουσίες πολύ υψηλής ανησυχίας και παράλληλα έχουμε τον κανονισμό βιοκτώνων και ε, ζυζανιοκτώνων. Και μπορεί να το ακούσατε και πέρυσι, όπου είχαμε μια ολόκληρη ιστορία για τα κριτήρια. Τώρα τα κριτήρια αυτά έχουν υιοθετηθεί, έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Βασικά τι σημαίνει αυτό. Έχουμε παράλληλα συστήματα για εντοπισμό του προβλήματος. Οπότε είναι πρόβλημα αυτό γιατί μπορεί εκεί να υπάρχουν ε, κάποιες αναντιστοιχίες και <clears throat> στη φάση της διαχείρισης του προβλήματος βλέπουμε στα δεξιά για κάποιες νομοθεσίες όπως στα καλλιτικά και στα παιχνίδια υπάρχει κάτι το οποίο απαγορεύει τις καρκινογόνες ουσίες αλλά δεν υπάρχει τίποτα για τους ενδοκρινικούς διαταράχτες και υπάρχουν και άλλες, ε, και άλλες, και άλλες λεπτομέρειες που δεν έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε αυτή τη στιγμή γιατί μου δώσατε μόνο 10 λεπτά. Στο ΡΙΤΣ ε, ο εντοπισμός ε, των ενδοκρινικών διαταρακτών ως ουσίες πολύ ψηλής ανησυχίας ε, για να φτάσουμε στον αναγνώριση και στο χαρακτηρισμό της ουσίας παίρνει πολύ χρόνο, αλλά δεν σημαίνει αυτόματα και απαγόρευση της χρήσης, για παράδειγμα, από τις φενόλες που έχουν εντοπιστεί ως ενδοκρινικοί διαταράκτες. Δύο έχουν απαγορευτεί τελείω. Από το 2021 όμως θα αρχίσει αυτό, ε, ενώ έχουν αναγνωριστεί ως διαταράκτες από το 2012 και από το 2013 κάποιες άλλες. Παίρνει πολύ χρόνο λοιπόν ο έλεγχος, η αναγνώριση, η ταυτοποίηση και η απαγόρευση. It's very sensitive. Uh, <laughs> oh. Yeah, so to conclude, uh, this is the, in, in a nutshell, the regulatory needs still uh, for endocrine disruption. Έχουμε λοιπόν ε, ανάγκες για νομοθεσία, έχουμε ανάγκη για εναρμόνιση και οριζόντια προσέγγιση για τον εντοπισμό και αναγνώριση αυτών των χημικών και έπειτα για τη διαχείριση του προβλήματος πρέπει να ε, καλύψουμε τα μεγάλα και πολυάριθμα κενά. Και να επιταχύνουμε βέβαια και όλη τη διαδικασία. Και αυτό είναι σύμφωνο με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον Μέχρι το τέλος του 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια στρατηγική για μη τοξικό περιβάλλον ώστε να εξασφαλίσει συγκεκριμένα την ελαχιστοποίηση έκθεση στου ενδοκρινικού διαταράχτες. Μέχρι το 2020 να έχει εναρμονίσει κριτήρια με τη βάση του κινδύνου για τον εντοπισμό των διαταρακτών και όλε αυτέ οι ουσίε θα πρέπει να τοποθετηθούν στους υποψήφιους, στον κατάλογο υποψηφίων για ένταξη στο ΡΙΤΣ και όπως σας είπα έχουν εντοπιστεί μόνο 12 χημικά από γύρω στα 120. Πολύ ωραία θα ήταν μόνο 12 να είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες, αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ. Φυσικά κάτι τέτοιο παίρνει ε, ε, χρόνο και χρήμα, ειδικά από την πλευρά της Επιτροπής, αλλά η Κομισιόν Προσπαθεί να περικόψει την γραφειοκρατία με την ατζέντα refit, αλλά πραγματικά θα θέλαμε να υπάρξει μεγαλύτερη δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου. Αυτά και αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ, είμαι στη διάθεσή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ερωταπαντήσεις θα γίνουν στο τέλος του πάνελ. Και τώρα το λόγο θα πάρει η κυρία Τσιγκώτη για να κάνετε δική της παρουσίαση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ε, ευχαριστούμε που οργανώσετε αυτή την ακρόαση. Είμαι η Νατάσα Τσινκόντι Είμαστε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που εργαζόμαστε σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος, health and και έχουμε συνεργασία με ομάδες περιβαλλοντικές ε, και εκπροσώπου της χημίας, του τομέα υγείας και ερευνητικά κέντρα. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. για τους ε, διαταράκτες, τους ενδοκρινικούς. Έχουμε πολλές φορές κάνει συζητήσεις. Σήμερα θα εστιαστώ στον τρόπο με τον οποίο η παρούσα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το, ε, στο παρόντα της κανονισμό η Επιτροπή ασχολείται με ένα θέμα το οποίο για τη δημόσια υγεία είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να είμαστε το καλύτερο, όσο καλύτερο γίνεται. Λοιπόν, Κοίτα. λοιπόν για να μπω σε λεπτομέρειες. Δεν θα σας ε, μιλήσω παρά από την πλευρά της δημόσιας υγείας. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι διαταράκτες αυτοί είναι παντού, είμαστε εκτεθειμένοι καθημερινά και αυτό το οποίο βλέπουμε αφενός είναι ότι οι επιστημονικές μελέτες και τα πορίσματα συνδέουν την έκθεσή μας με χημικές ουσίες και με την ε, παρουσία διαφόρων νοσημάτων, χρόνιες ασθένειες, καρκίνους, κάποιες ασθένειες που έχει κανείς όλη του τη ζωή οφείλονται σε αυτούς τους διαταράκτες. Ακόμη και σε θέματα αναπαραγωγής υπάρχει πρόβλημα. Και αυτή η αξιολόγηση κάτι το οποίο οδήγησε και τους υπεύθυνους δημόσιας υγείας στο να θέλουν να συμμετάσχουν στο όλο εγχείρημα. Ξέρουμε ότι έχει γίνει από την ε, ε Διεθνείς από την ε, Διεθνή Ομοσπονδία Γυναικολόγων και άλλους ε, ονώσεις που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία, ότι θα πρέπει να υπάρξει η σχετικός κανονισμός για τους ενδοκρινείς διαταράκτες ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την ε, επιδείνωση της κατάστασης και να προστατεύσουμε τους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει η κατάλληλη πρόληψη και να υπάρξουν οι κατάλληλοι κανόνες ώστε να, δυνητικά να προστατεύσουμε τους πολίτες. Βεβαίως ξέρουμε ότι υπάρχει και το ε, οικονομικό κόστος για τα διάφορα συστήματα δημόσιας υγείας και θα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε τις καλύτερες έρευνες και μελέτες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο κοστίζει πάρα πολλά εκατομμύρια ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν χημικές ουσίες οι οποίες ευθύνονται ε, για τέτοιου είδους θέματα όπως οι δυσφενόλοι, ε, ουσίες που περιέχονται στα εντομοκτώνα και αναφέρω αυτούς τους ρυθμούς διότι αυτό αυτό το οποίο έχουμε σήμερα είναι μόνο η εικόνα της κορυφής του παγόβουνου. Όταν λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός, πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε οι σχετικές οδηγίες και κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι καλύτερα, διότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι το επαρκές τα κριτήρια για τα βιοκτώνα και τα εντομοκτώνα, όπως ξέρετε, ε, έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ να θεσπιστούν. Ξέρουμε ότι υπάρχει Σουηδία η οποία έχει προσφύγει κατά της καθυστέρησης αυτή και πιστεύουμε ότι το βάρος της απόδειξης είναι πάρα πολύ υψηλό και φαντάζομαι ότι αυτό πρέπει να γίνει μέρος όλων μας. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ένα συνοδευτικό έγγραφο ε, σε όλες αυτά τα ε, επίσημα έγγραφα για να καταλαβαίνει κανείς περί τίνος πρόκειται. Από τη δική μας άποψη λοιπόν πρέπει να σας πω ότι η δυσφενόλη α είναι μία από τις ε, ουσίες που ενέχονται για περισσότερο από άλλες για τις ενδοκρινικούς διαταράκτες. Γνωρίζουμε πάρα πολλά ε, στοιχεία για το θέμα αυτό και ξέρουμε ότι πολλές ε, φορές πίσω από τις διάφορες επιστημονικές αποφάσεις και αποτελέσματα κρύβονται και διάφοροι πολιτικές για να διαμορφωθούν οι κανονισμοί. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα η έκθεση των πολιτών είναι πολύπλευρη, έχουμε τέτοιου είδους ουσίες στα καλλιντικά, στα παιχνίδια. Και ολοκληρώνοντας, προσπαθώντας να κάνουμε συστάσεις για περαιτέρω δράση, πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για τα κριτήρια που αφορούν τα εντομοκτώνα και τα βιοκτώνα, ώστε να δώσουμε κάποιες οδηγίες για το πώς μπορεί κανείς να προστατευτεί. Ξέρουμε ότι στην οδηγία REACH συμπεριλαμβάνονται κάποια στοιχεία για τους διαταράκτες αυτούς, αλλά θα πρέπει να γίνουν περισσότερα, θα πρέπει να ταυτοποιηθούν περισσότερες ουσίες. Εάν δεν μπορεί να το κάνει από μόνο της για να βελτιώσει την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να στραφεί προς τα κάτι μέλη τα οποία έχουν περαιτέρω προωθήσει τις έρευνες τους, τη Δανία, η Γαλλία, ώστε να δουν πώς ε, ε, διαμορφώνεται η δική τους στρατηγική. Στην ε, Γαλλία αύριο θα ψηφίσει η Γερουσία μια στρατηγική βάση των 70 περίπου μέτρων για την βελτίωση της οδηγίας. Ευχαριστώ. Σας, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριος Πέτερ Κόριταρ από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΝΒΙ, παρακαλώ, Γενικής Περιβάλλοντος. Έχετε το λόγο. Να έχουμε ετοιμάσει και μια παρουσίαση, σύντομη. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε και μας ε, χώρο και βήμα εδώ να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας. Θα ήθελα καταρχάς να σας ε, δώσω το ιστορικό. Ποιες είναι οι πολιτικές ε, της Ένωσης στον τομέα ε, των ενδοκρινικών διδακτών. Πώς ξεκίνησαν ουσιαστικά τα πράγματα. Ξεκίνησαν κάπου το 1996. Οπότε και δημοσιεύτηκε ένα βιβλίο από την κυρία Κόμπερν. Το κλεμμένο μας μέλλον, Our Stolen Future, όπου εκεί μιλά για την ε, επίπτωση κάποιων πρακτικών ε, στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Αυτό ήταν ένα βιβλίο που διαβάστηκε από πάρα πολλούς και ε, δημιούργησε πολλέ συζητήσει. Οδήγησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κατέληξε κάποια συμπεράσματα το 1998, που ζητάει μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσει η Κομισιόν το ζήτημα των αντιπρών διαταρακτών αλλά προληπτικά μέτρα και να πει πώ θα προχωρήσει. Και η Κομισιόν ε, υιοθέτησε μια στρατηγική το 1999 για του ανθρωπινικού διαταράκτε, που μέχρι σήμερα ε, ουσιαστικά είναι η στρατηγική που έχουμε σε κοινωτικό επίπεδο για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά την πολιτική μας. Δεν ε, περιγράφεται αυτό τόσο σε αυτή τη στρατηγική που προανέφερα, αλλά στο δρόμο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον. Στόχος λοιπόν είναι η ελαχιστοποίηση της έκθεσης στους ανακρινικούς διαταράκτες, στον εντοπισμό ορισμένων δράσεων μέχρι το 2020 για την ταυτοποίηση των ουσιών αυτών και την ενίσχυση των μέτρων. Πού είμαστε σήμερα σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των ενδοκρινικών διαταρακτών. Σε όλα τα νομοθετήματα ρυθμίζουμε του ε, ενδοκρινικού διαταράκτε, εφόσον πρόκειται για κάποιο νομοθέτημα που ρυθμίζει τα χημικά, τι χημικέ ουσίε. Δεν ε, το έχουμε δηλαδή παραγνωρίσει το θέμα αυτό. ταλεντικά, παιχνίδια. Υπάρχουν και συγκεκριμένα νομοθετήματα με ειδικέ διατάξει για του αναπτυνικούς διατάξει από το 2000 και μετά, που είχαμε δηλαδή την οδηγία για τα για παράδειγμα. Είπαμε ότι μπορεί αυτέ οι ουσίε να είναι <clears throat> ουσίε προτεραιότητα και οι εκπομπέ στο περιβάλλον αυτών των ζώων θα πρέπει ε, να εξαλειφθούν. Στο ΡΙΤΣ έχουμε ειδική διάταξη επίσης λέμε ότι μας ανησυχούν οι ουσίες αυτές και ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ε, έγκρισης άδεια. Επίσης, ε, στον κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά και για τα βιοκτώνα, Έχουμε πολύ ε, αυστηρές εκεί διατάξεις. Λέμε ότι οι ενδοκρινικοί διατάξεις θα πρέπει να αδειοδοτηθούν για χρήση σε προϊόντα βιοκτώνα ή φυτοπροστατευτικά. Τέλος, το 2017 τελευταίο νομοθέτημα, ο κανονισμός για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Έχουμε και μια νέα πρόταση, επιτάπητος, οδηγία για το πόσιμο νερό. Ε, προτείνουμε ένα παράρτημα της εν λόγω οδηγίας να τροποποιηθεί και να προσθεθούν τρεις μεμονωμένες χημικές ουσίες που έχουν ε, ε, ιδιότητες διαταραχής του ανδοκρινικού συστήματος για να σας ενημερώσω για το τι κάνουμε τώρα. Ολοκληρώνουμε το έργο για τα κριτήρια για τους ολοκληρικούς διαταράκτες ε, στον κανονισμό για τα βιοκτώνα και τα ε, φυτοφάρμακα. Ήδη από την 7η ε, Ιουνίου ισχύουν, ενώ στην άλλη περίπτωση είμαστε στην μάλλον για τα βιοκτώνα θα ισχύσουν από την 7η Ιουνίου του 2018 και για τα ε, φυτοφάρμακα ακόμα συνεχίζεται ο έλεγχος Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, μάλλον θα εγκριθούν από τον Νοέμβριο του 2018. Νομοθεσία, νέα επιστημονικά κριτήρια. Πρέπει για να θεωρήσουμε ότι μια ουσία προκαλεί ενδοκρινική διαδίκτυα, θα πρέπει να προκαλεί μια ε, επίπτωση. Πρέπει να αποδεχθεί η σχέση αιτίου-αιτιατού. Αιτίου και ένα συσχετισμό μεταξύ αυτών των δύο, τη ενδοκρινική δράση και τη ανεπιθύμητη ενέργεια. Και μελετάμε όλε τι διαθέσιμε επιστημονικέ πληροφορίε. Δεν υπάρχει μια νέα δοκιμή ή μελέτη που θα μας πει αν μια ουσία είναι ε, υπεύθυνη για αναπληκτικές διαταρχές ή όχι. Πρέπει να γίνουν πολλές ε, μελέτες ταυτόχρονα. Παράλληλα τώρα με την ε, εκπόνηση των κριτηριών έχουμε ξεκινήσει και τη συγγραφή ενός ε, κειμένου κατευθυντηρίων γραμμών. Ζητήσαμε από την ΕΦΣΑ και τον ΕΚΑ να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές Έγινε για το πρώτο σχέδιο των κατευθυντήρων γραμμών μια δημόσια διαβούλευση. Οργανώθηκε και ένα εργαστήριο με τα κράτη-μέλη που είδαμε ε, αν ε, είναι ε, τα αυτά τα κριτήρια και ελπίζουμε το τελικό έγγραφο να είναι έτοιμο μέχρι τα μέσα του τρέχοντος έτους. Πέραν του έργου μας από των κριτηρίων για τους ανδροκρινικούς διαταράκτες, προχωρούμε και σε ό,τι αφορά τις κατευθύνσεις γραμμές για τις δοκιμές για τις μελέτες. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για το ενταυτοποίηση των ενδοκρινικών διαταρακτών. Ξεκίνησε το έργο αυτό ήδη από το 1999 2000 Στο πλαίσιο του ΟΣΑΚ έχουμε μέχρι στιγμή 13 τέτοιες κατευθυντήριες γράμμες για ταυτοποίηση τέτοιων οργανισμών για την αναγνώριση ιδιωτήτων ε, ενδοκρινικής διαταραχής. Επίσης υπάρχει και ένα έγγραφο καθοδήγησης για το πώς θα ερμηνεύονται τα αποτελέσματα των δοκιμών και μελετών. Υπάρχουν βέβαια ακόμη ε, κενά και λήψεις. Πολλές μελέτες το καταδεικνύουν αυτό. Είχαμε και μια έκθεση του Ισπακόσμου Οργάνωσης Υγείας το 2013, τη γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ Επίσης, από το 2013. Έχουμε και δικέ μας μελέτες που λένε ότι υπάρχουν κενά ακόμα, γι' αυτό ξεκινήσαμε λοιπόν τις προσπάθειες ε, να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των καθεντήριων γραμμών για τις δοκιμές και έχουμε αναθέσει διάφορες μελέτες ε, Παραδείγματο χάρη για τη διαταραχή του, τον, ε, θηροειδική, είχαμε ένα εργαστήριο και είδαμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. για το retinoid signaling pathway και θα έχουμε και σύντομα μια έκθεση για την άρχιση προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων δοκιμών. Και όταν έχουμε εντοπίσει όλα τα κενά, θα πρέπει να δούμε τι είναι το πιο επίγον, πού πρέπει να διαθέσουμε ε, πόρους και προσπάθειες σε λίγες εβδομάδες θα την έχουμε αυτήν την ε, μελέτη. Θέλουμε να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο όμως ε, για τη θεωρητική διαταραχή το κοινό Κέντρο Ερευνών προσπαθεί να βελτιώσει τις in μεθόδους Επίσης και για τις ε, δοκιμές in vivo προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά ε, και να βελτιώσουμε τις δοκιμές σε ό,τι αφορά πάντα τη θεωρητική διαταραχή. Επίσης προκηρύξαμε ένα διαγωνισμό για μάλλον πρόσκληση υποβολής 5 ε, εκατομμύρια ευρώ εν το ποσό που θα διαθέσουμε για ένα project για την ανάπτυξη δοκιμών για τους διαταράκτε διαταράκτες. 18 Απριλίου λίγη προθεσμία και ελπίζουμε τα επόμενα 3-4 χρόνια να έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοριτάρ. Έχουμε εκπροσώπους και από την ε, Γενική Διεύθυνση Υγείας, τον κύριο Μπέραντ, την, την κυρία Μίστεν και τον Τζόναθαν Μπριν. Θα ήθελα να σας ερωτήσω εάν Θέλετε εκ μέρους Γενικής Διεύθυνσης Υγείας να λάβετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όχι, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτε άλλο, δεδομένου ότι ο, ο, ο κύριος Κόριταρ σας εξέθεσε τα θέματα ε, τα δικά μας και έχουμε ε, συντονιστεί μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Επίσης με ενημερώνουν και ότι η DG Ανάπτυξης έχει στείλει εδώ τον κύριο Στρέκ και τον κύριο Φόγερσαν. Θα ήθελα να τους ερωτήσω επίσης εάν θέλουν να λάβουν το λόγο, να κάνουν κάποια παρατήρηση. Καλημέρα σας. Είμαι ο Γεωργ Στέφεν, ο συνάδελφος Γιούργεν Φόλγκεστεν δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σήμερα. Τον, εγώ εκπροσωπώ τη Γενική μου Διεύθυνση και δεν έχω προς το παρόν να κάνω καμία παρατήρηση. Όπως είπε και ο συνάδελφος, μας κάλυψε η παρουσίαση του κυρίου Κόριτο. Ευχαριστώ. Εάν υπάρξουν ε, ερωτήσεις, ενδεχομένως μπορείτε να απαντήσετε. Αυτή τη στιγμή Συνάδελφοι, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, κύριος Πίτερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέσσερα θέματα έχω σημειώσει για τα οποία θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. δεν συμφωνούμε με κάποια από τα βήματα τα οποία ακολούθησε η Κομισιό σε θέματα πραγματογνωμοσύνης, ε, ε, ταχύτητας. Ακολουθήσαμε τα λάθος πορίσματα. Το θέμα δεν είναι ποιος είναι ένοχος και ποιος δεν έχει αυτή την υπόθεση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες ήδη το έχουν μελετήσει το θέμα και Ξέρουμε ότι είναι επικίνδυνες ε, είναι επικίνδυνοι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Μια άλλη ερώτηση. Η καφεΐνη είναι επικίνδυνη, διότι όντως επηρεάζει τις ορμόνες. Κάποιοι λένε, μα πιείτε 20 φλιτζάνια καφέ, θα πάθετε κάτι. Εγώ δεν πίνω 20 φλιτζάνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν παίρνονται κάποιες ε, αποφάσεις, αλλά θα πρέπει πάντα να βλέπουμε και ποια είναι η προσλαμβανόμενη δόση κάποιου προϊόντος. Και σωστά λέτε ότι θα πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση ανάλογα με την που χρησιμοποιούνται ε, αυτές οι ουσίες. Ε, Φερρυπίν, στα παιχνίδια ή σε ιατρικά εργαλεία και σε ιατρικό εξοπλισμό. Είναι διαφορετική η χρήση τους. Αν πρέπει ένας γιατρός να γλιτώσει τη ζωή ενός ασθενούς, μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους ουσίες οι οποίες ενδεχομένως περιέχονται στα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει. Επίσης, υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών που, των ε, διαταρακτών που χρησιμοποιούνται στα εντομοκτώνα, στα ζυζανιοκτώνα και στα καλλιντικά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ των φυτοφαρμακευτικών προϊόντων, των καλλιντικών και των ε, φυτοφαρμάκων. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία είναι όντως επικίνδυνα. Και σίγουρα υπάρχει επηρεασμός ε, και της επιστήμης και της πολιτικής Για τα καλλιντικά, παραδείγματο χάρη, θα έχουμε μεγαλύτερα ε, προβλήματα αν ο κόσμος ε, θεωρεί ότι γίνεται πιο όμορφο με τη χρήση των καλλιντικών. Το τρίτο, συμφωνείτε ότι δεν θα πρέπει να διαφοροποιούμε πολύ τα πράγματα. Αν δηλαδή ε, συλλάβουμε ένα σύστημα, σχεδιάσουμε ένα σύστημα, θα πρέπει Σίγουρα να κάνουμε βέβαια τη διάκριση μεταξύ ε, παιχνιδιών ε, και χημικών ουσιών, αλλά όχι να διακρίνουμε τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται τα σακάλι δικά από αυτές που χρησιμοποιούνται κάπου αλλού. Είπα για την πολιτική και την επιστήμη. Εμείς έχουμε το δύσκολο καθήκον να ε, μεταφέρουμε τις επιστημονικές ενδείξεις σε πολιτική, σε νομοθεσία και σίγουρα Ε, ξέρετε ότι υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα με την ε, γλυφοσάτη, όπου εκεί έχουμε μια διαφορά μεταξύ της κοινωνικής αντίληψης και των επιστημονικών ε, απόψεων. Θα πρέπει κατά την άποψή μου να έχουμε ένα λογικό σύστημα κατανοητό, μια ευρωπαϊκή στρατηγική συνεκτική είπε κάποιος, καλό είναι αυτό. και δεν ξέρω αν τώρα που είμαστε στην αρχή θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για εξαιρέσεις. Ε, Thanks a lot, Chair, and thank you to all the speakers and σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και περισσότερο ακόμα τους ε, εισηγητές μας, ε, ε, τους προσκεκλημένους μας. Κατανοώ το η σημασία αυτού του θέματος και γι' αυτό και το συζητάμε σήμερα, γιατί και πάλι διαπιστώνουμε την πολύ μεγάλη ανησυχία των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις χημικές ουσίες που επηρεάζουν τη λειτουργία των, των ενδοκρινών αδένων. Για να νομοθετήσουμε για ισχυρότερη η προστασία από τις ουσίες αυτές ε, είναι πολύ δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι πολύ περισσότερη και σημαντική δουλειά ε, έχουμε ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να πω ότι είναι θετικό που η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της να προβλέψει κριτήρια στα βιοκτώνα και στα ζυζανιοκτώνα. Αυτό είναι ένα πρώτο καλό βήμα, αλλά για τους πολίτε μας και για το περιβάλλον πιστεύω στεναρά πως χρειάζεται κριτήρια όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά είναι κάτι το οποίο θα παραμένει σταθερό στα αιτήματα ε, για οριζόντια κριτήρια. Αυτό θέλω να τονίσω. Δεν είναι θέμα αναγνώρισης δύο συγκεκριμένων ειδών προϊόντων, αλλά εμείς ως σοσιαλιστές και δημοκράτες παραμένουμε σταθεροί στην στην, στο έτοιμά μας ότι χρειαζόμαστε οριζόντια κριτήρια ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να προστατεύονται από όλους, όλες αυτές τις χημικές ουσίες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να ασκούμε πίεση ε, σε αυτό το τομέα και αναμένουμε ε, οι ουσίες αυτές να παγορευτούν στις συσκευασίες για τα τρόφιμα, στα παιχνίδια και στα καλλιτικά ε, και για να υπάρξει αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση και συγκεκριμένη δράση από την Κομισιόν. Γιατί η αδράνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα οδηγήσει σε κατάσταση όπου θα έχουμε μεμονωμένα κρατημέλη να αναλαμβάνουν μεμονωμένες δράσεις. Πιστεύω πως μακροπρόθεσμα Εάν έχουμε διαφορετικά πρότυπα στα διάφορα κράτη θα είναι πιο δύσκολη κατάσταση για όλους. Ούτε για τους καταναλωτές που δεν θα ξέρουν τι επίπεδο προστασίας δεν αμένουν, αλλά θα είναι και δύσκολο για τους παραγωγούς που θα υποφέρουν από τα αποκλίνοντα πρότυπα. Και έχω και κάποιες ερωτήσεις Άκουσα την παρουσίαση της Κομισιόν που υποτίθεται ότι ε, εργάζεται για μια νέα στρατηγική για ελαχιστοποίηση της έκθεσης στους, ε, στις χημικές ουσίες αλλά και έχει δώσει και νέα εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα φέτος και θα ήθελα να γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει με τη στρατηγική και πότε θα δημοσιευτεί. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω από τους ε, ομιλητές μας τι πιστεύουν για την δράση της Κομισιόν και αν την βρίσκουν ικανοποιητική ως φιλοδοξία και από την άποψη του επιστημονικού πεδίου και τέλος για την ΕΚΑ. Η Κομισιόν εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια για να τα ε, ελέγξει αν οι ουσίε μπορούν να μπουν στην αγορά ή όχι, αλλά πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση και σε κάποια πρώιμα στάδια. Ορισμένοι επιστήμονε ε, ε, υποστηρίζουν ότι κάποιες ε, τοξικέ δοκιμέ πριν από το τρίτο επίπεδο δεν είναι επαρκή και μπορεί εύκολα κανεί να τα χειραγωγήσει τα στοιχεία οπότε θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σα γνώμη και θα θέλαμε να ξέρουμε και περισσότερα στοιχεία για τι αρχικέ διαδικασίε. Σα ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ροζιέρης. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με εκπλήσουν κάποια θέματα τα οποία άκουσα από τους συναδέλφους. Πρέπει να πω ότι είμαστε από την δεκαετία του 70 ενήμεροι, διότι υπήρχαν επιστημονικές ε, ε, ενδείξεις και μαρτυρίες για τα θέματα αυτά. Δεν είναι θέμα πολιτικής άποψης. Έχουμε αποδείξεις από την επιστημονική κοινότητα εδώ και περισσότερο από 40 χρόνια. Ξέρουμε επίσης ότι υπήρξε και καταδίκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάποια θέματα. Τα γεγονότα είναι γνωστά σε όλους. Και Γι' αυτό και κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει, που ζητά να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτούν οι πολίτες της Ευρώπης. Πρόκειται για σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας και εμείς ως εκπρόσωποι των πολιτών έχουμε την ευθύνη να προωθήσουμε τα πράγματα και να θέσουμε πρώτων ευθυνών τους αυτούς οι οποίοι ενέχονται σε αυτή την υπόθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ούτως ή άλλως τους και τις παρεμβαίνοντες, παρεμβαίνουσες για το θέμα αυτό. και Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να βοηθήσουμε την Επιτροπή όλοι ώστε να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις, το καλύτερο δυνατό πλαίσιο. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ποια είναι η καλύτερη ανταπόκριση ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Δεν είναι θέμα υποκειμενικό όσον αφορά τα διάφορα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ε, ασφαλή χρήση όλων αυτών των ενεχόμενων προϊόντων και ουσιών υπέρ των πολιτών της Ευρώπης και γι' αυτό προσπαθούμε να κατευθύνουμε έτσι τα πράγματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία που είναι, ήταν εξαιρετική και ευχαριστώ για την ποιότητα των παρεμβάσεων. Ακόμα όμως έχω αμφιβολίες ε, σε σχέση με την πραγματική φιλοδοξία της ε, Κομισιόν που αργεί να ασχοληθεί σοβαρά Ειδικά σε μια τέτοια φάση όπου οι πολίτες ε, μας ζητούν να ενδιαφερθούμε για αυτό το πρόβλημα και ο επιστημονικός κόσμος. Εγώ πραγματικά βρίσκομαι σε μια κατάσταση που ενώ ο, δηλαδή ο γιατρός ε, σπουδάζει, ο ασθενής ε, μπορεί να πεθάνει. Έτσι αισθάνομαι. Εγώ ανέκαθεν ναι, να έχω ενδιαφερθεί για αυτό το θέμα από την αρχή της θητείας μου με διάφορους συναδέλφους, ιδιαίτερα με τον Πάβελ, με τον οποίο ε, συμφωνούμε και έχει, έχουμε υποβάλει και προφορική ερώτηση από το 2015, την οποία στηρίξαν πολλοί συνάδελφοι και ρωτήσαμε τότε Ζητήσαμε από την Κομισιόν να υιοθετήσει επιστημονικά κριτήρια για τις ε, ουσίες αυτές, για τα βιοκτώνα και τα ε, ζυζανιοκτώνα ε, και τον Οκτώβριο πέρυσι απορρίψαμε την πρόταση της Κομισιόν που είχε ορίσει, είχε προτείνει μάλλον κοινά επιστημονικά κριτήρια για αυτές τις για αυτές τις ουσίες. Εμείς θεωρήσαμε πως δεν ήταν αποδεκτό το να εξαιρεθούν κάποιες ουσίες καθώς έλειπε και ο ορισμός των υπόπτων μορίων. Ε, πριν από λίγους μήνες στείλαμε μια νέα ερώτηση προφορική για μια, και ζητήσαμε μια νέα στρατηγική για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες ώστε να μειωθεί στο μήνυμο η έκθεση των Ευρωπαίων πολιτών σε αυτές τις ουσίες πέρα από τα βιοκτώνα και τα ζυζανιοκτώνα. Και αυτό για να πω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα που εμπλέκονται και δεν επικρατεί απόλυτη ε, διαφάνεια. Αυτή είναι η απόψή μου, αλλά... Κάτι που είναι σαφές, είναι σίγουρο, είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κάνει εκπτώσεις ε, εφόσον ε, πρόκειται για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Να μιλήσω ωστόσο για μια πτυχή που μέχρι στιγμής δεν την έχουμε αντιμετωπίσει επαρκώς τις οδηγίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί την έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράχτες ως ένα πρόβλημα αντίστοιχο με αυτές αυτό της κατηγορίας ουσιών που είναι προβληματικές όπως οι καρκινογόνες. Ε, κατά συνέπεια, οι ουσίες που εντοπίζονται και αναγνωρίζονται ως ενδοκρινικοί διαταράχτες θα πρέπει να απαγορευτούν και να αντικατασταθούν από άλλες ουσίες πιο ασφαλείς. Η εμπειρία από το contaminants όμως μας δείχνει ότι οι πιο σοβαροί ενδοκρινικοί διδρακτές μπορεί να μην ενταχθούν εκεί. Legacy contaminants λέγονται αυτές οι ουσίες που μένουν στο περιβάλλον ε, πολύ μετά από την παραγωγή τους και τη χρήση τους, ακόμα και αν αυτή έχει απογορευθεί. Οι legacy contaminants είναι συσσωρευτές που σωρεύονται σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και άρα ε, τίθεται το θέμα της ασφάλειας ε, των τροφίμων, PCB, η... Ε, διάφορα πυρήμαχα υλικά, ε, μπορεί να βρεθούν λοιπόν τέτοια μικροσωματίδια και μέσα στο νερό και μπορεί να μένουν για πολλά χρόνια ενεργές αυτές οι ουσίες. Τώρα στην παραγωγή της γεωργίας μπορεί και τα ζώα να ε, σωρεύουν ε, ενδοκρινικούς διαταράχτες, τοξικές ουσίες που υπάρχουν στους βοσκότοπους θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια συγκεκριμένη στρατηγική ώστε να προστατευτεί μια σωστή γεωργική δραστηριότητα, κτηνοτροφική βασικά δραστηριότητα στις ε, μολυσμένες περιοχές. Να εντοπιστούν δηλαδή εναλλακτικέ πηγές ε, ζωοτροφών για τα ζώα και θα μπορούσε θα, θα έπρεπε μάλλον η γεωργική παραγωγή να μην υπόκειται τόσο σε αυτή την βιοσόρευση. Ε, εκτός δηλαδή από την απέτηση για άμεση, πάυση, απαγόρευση στρατηγική της Κομισιόν η οποία να είναι φιλόδοξη, τόσο φιλόδοξη όσο και σημαντικό είναι αυτό το θέμα, θα ήθελα να είμαστε πιο ρεαλιστές και να καταλάβουμε ότι ενώ βελτιώνουμε τη βιωσιμότητα των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούμε, θα αντιμετωπίσουμε και τις, τις νέες περιβαλλοντικές ε, κληρονομιές. Οι αυριανοί πολίτες δηλαδή που γεννιούνται τώρα θα υποστούν τις συνέπειες των όσων εμείς κάνουμε και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καν σε θέση να φανταστούμε ε, πώς θα εμποδίσουμε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιράντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους εισηγητές σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ακρόαση που προκαλεί το ενδιαφέρον την κοινή γνώμη, αλλά κυρίως κάτι το οποίο αφορά κυρίως τους καταναλωτές και θα ήθελα την κυρία Θαμπότη να ερωτήσω πώς έχει η ενημέρωση για τέτοιου είδους ουσίες. Επίσης είπαμε ότι υπάρχει ένα ε, πρόβλημα μεγάλο για το περιβάλλον, για τη δημόσια υγεία, οικονομικό, γιατί έχουμε προστιθέμενα προβλήματα υγείας. Η Επιτροπή κάτω από την πίεση που δέχθηκε, χρειάστηκε πριν από τις 2013 να κάνει κάποιες ρυθμίσεις για αυτές τις ε, πολύ επικίνδυνες ουσίες. Έκανε όμως, όπως είπαν οι επικρίσεις τότε, κάτι το πάρα πολύ αφηρημένο. Διότι πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με ένα κοκτέιλ ορμονών και ουσιών που είναι επιβλαβείς. Ξέρουμε επίσης ότι χρειάστηκε να κάνει ε, κάτι από το 2013 και μετά η Κομισιό κάτω από πιέσεις και από την βιομηχανία και πέρασε το θέμα αυτό από την ε, μία γενική διεύθυνση στην άλλη και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή Γιούνκερ άλλαξε τον προσανατολισμό του θέματος και το ποιες ουσίες θα συμπεριλαμβάνονται το δεδομένο ότι είμαστε όμως σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να έχει ένα υποχρεωτικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει όλοι να ακολουθούμε ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις ανάλογα με το ποιο κράτος βρίσκεστε για την απαγόρευση αυτών των ουσιών. Έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα ανισότητας αντιμετώπισης ενός σημαντικού προβλήματος δημόσιας υγείας για τους πολίτες μας. Τι, έχουμε, λοιπόν, τι έχετε λοιπόν να μας πείτε για την ε, δημόσια υγεία, για, για, γιατί μιλήσατε κυρία Τσινκώτη για 156 εκατομμύρια ευρώ κόστος. Ε, τι έχετε λοιπόν να μας πείτε για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος βουλευτής το λόγο. Οπότε ίσως είναι τώρα ώρα να ακούσουμε σε δύο γύρους τις απαντήσεις. Πρώτα αν θέλουν οι εκπρόσωποι της Κομισιόν και μετά τα μέλη του πάνελ. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω και να σχολιάσω ορισμένα από αυτά που υπόθηκαν, ιδίω σε σχέση με τα κριτήρια που έχει εγκρίνει η Κομισιόν. Για τα φυτοπροστατευτικά πρέπει και για τα βιοκτώνα. Νομίζω ότι πολλοί βουλευτές είπαν ότι είναι μεγάλη αυτή η ιστορία, μίλησαν για τις καθυστερήσεις και για το γεγονός ότι υπήρξε και απόφαση του δικαστήριου που καταδίκασε την Κομισιόν που δεν είχε αναλάβει έγκαιρα δράση. Πολλές φορές σας έχουμε δώσει εξηγήσεις για το θέμα αυτό, ιδίως όταν είχαμε συζητήσει το σχέδιο κριτήριων στο Επιτροπεριβάλλοντος εδώ στο Κοινοβούλιο. Ένα από του λόγου είναι κάτι που ισχύει και σήμερα, οι διαφωνίε μεταξύ επιστημόνων, κάτι που δυσκολεύει και την Κομισιόν να καταλήξει σε προτάσει για τα κριτήρια. Το Κοινοβούλιο δεν είχε κάνει δεκτά τα κριτήρια που πρότεινε η Κομισιόν για τα ζυζανιοκτώνα, όχι όμως λόγω του επιστημονικού περιεχομένου, αλλά αποκλειστικά και μόνο για μία ρήτρα που αναφερόταν συγκεκριμένα σε ουσίες που ρυθμίζουν ε, αυξητικούς παράγοντες για τα φυτά που μπορεί να είναι και διαταράκτες. Ό,τι αφορά τα βιοκτώνα έχουμε, όπως πάμε τα κριτήρια και έχουμε και για τα ζανιοκτώνα ένα έγγραφο το οποίο μελετάται αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο και βέβαια ε, μετά θα το εγκρίνει και το Συμβούλιο. Εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι άτομα τα κριτήρια και δεν είναι αρκετά φιλόδοξα. Είπε ο Πέτερ Κόρτερ, ο συνάδελφος, αλλά και ο εκπρόσωπος του ΕΚΑ ότι έχουν ταυτοποιηθεί ουσίες που υποπτευόμαστε ή γνωρίζουμε ότι είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Και μπορούμε να δούμε όλα τα επιστημονικά δεδομένα και τα διάφορα άλλα στοιχεία που υπάρχουν. Άρα η Κομισιόν θεωρεί ότι έχει τα απαραίτητα μέσα στη διάθεσή της για να ταυτοποιήσει ενδοκρινικούς διαταράκτες. Κυρία Νταλή, νομίζω τώρα, μίλησε για οριζόντια κριτήρια. Η Κομισιόν πρέπει να σας πω, έχει προτείνει τα ίδια κριτήρια για τα ζανιοκτώνα και για τα βιοκτώνα. Γνωρίζοντα ότι οι ίδιε ουσίε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δύο διαφορετικέ κατηγορίε προϊόντων. Άρα ουσιαστικά αυτό ε, πηγαίνει προ κατεύθυνση του αιτήματο τη κυρία Ντάλη. Και ο εκπρόσωπο του ΕΚΑ επίση είπε για ταυτοποίηση των ε, ενδοκρινικών διατρακτών στο πλαίσιο του ΡΙΤΣ χρησιμοποιούμε και τον ορισμό τη Παγκόσμια Υγεία, που είναι βάση για τα κριτήρια που έχει προτείνει η Κομισιόν για βιοκτώνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική, η Κομισιόν πράγματι έχει ανακοινώσει πέρυσι τον Ιούλιο ότι θα εκπονήσει μια νέα στρατηγική με βάση την ίδια φυστάμενη που ισχύει από το 99, όπως είπε ο κ. Κότηρ. Κύριε Τσιγκώτη, είπε ότι είναι στα σερτάρια του Γενικού Γραμματέα. Δεν ισχύει αυτό. Αντίθετα, δουλεύουμε το κείμενο πριν 10 μέρε. Είχαμε μια διεπηρεσιακή συνάντηση για να δούμε την πρόοδο του έργου που συνεχίζεται. Αλλά δεν μπορώ να δεσμευτώ να σα δώσω μια συγκεκριμένη ημερομηνία, εφόσον ο Γενικό Γραμματέα είναι ο αρμόδιο. και συντονίζει όλε τι υπηρεσίε. Πάντω εργαζόμαστε επί του θέματο. Άρα αυτό που είπαμε το κάνουμε. Και είπε και ο κύριο Σκότηρ ότι με την ανακοίνωση θέλαμε να έχουμε περισσότερους πόρου για ερευνητικέ δραστηριότητε. Όπου να είναι θα διατεθούν αυτά τα κονδύλια. Και ένα τελευταίο σχόλιο για αυτό που ο κύριος Γιάρ για τη ρύθμιση των ουσιών με βάση την επικενδυνότητα και τον Hazard ή risk για διοκτώνα, ζενιοκτώνα είναι ξεκάθαρο. Οι επιστήμονε ότι θα πρέπει η απόφαση να λαμβάνεται με βάση την επικινδυνότητα, hazard. Το σέβεται η Κομισιόν. Σε άλλα νομοθετήματα η κατάσταση έχει... δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Το Σύνολο και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που εγκρίνουν όμω το γενικό κανονισμό πλαίσιο. Και αυτοί θα αποφασίσουν ακριβώ τι κριτήρια θα εφαρμόζονται. Ευχαριστώ. Ε, maybe... Δεν ξέρω αν θέλουν να αντιδράσουν στην αντίδραση της Κομισιόν κάποιοι συνάδελφοι. Αυτό μπορείτε να το κάνετε, αλλά μετά το δεύτερο πάνελ. Οι συνάδελφοι του πρώτου πάνελ, μήπως θα ήθελα να κάνουν κάποιες τελικές παρατηρήσεις. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Τα περισσότερα νομίζω απευθύνονταν στην Επιτροπή. Από την ΕΚΟ έγινε επίσης μια ερώτηση για τα τεστ ποιότητας για το ότιση. Έχουμε μια ομάδα η οποία κάνει αξιολογήσεις και ε, λέει στα κράτη-μέλη ποια είναι τα τεστ, ποιες είναι οι δοκιμές που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουν να ταυτοποιηθούν, να εντοπιστούν οι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Τι απαιτείται, λοιπόν. Αυτό αφορά τις δοκιμές, τα τεστ τα οποία μπορούν να μας δώσουν τις καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους διαταράκτες. Γενικά, για να επιταχυνθεί η διαδικασία, θα πω ότι η Επιτροπή πολύ πρόσφατα έκανε αναθεώρηση του ΡΙΤΣ και εντόπισε πολλές διαφορετικές δράσεις που θα μπορούσαν να αναλυφθούν από την ΕΚΟ και από άλλους για να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία, να επιταχυνθεί και η ΕΚΟ θα συνεργαστεί εκ του σύνεγγες με την Επιτροπή και άλλους φορείς ώστε να ε, προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο στάδιο στις απαραίτητες συστάσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμμετέχοντες, έτσι ολοκληρώθηκε η συζήτηση Πρώτο πάνελ. Εγώ είμαι από την ε, Σλοβακία και ο συνάδελφος από την Τσεχία. Σχεδόν είμαστε λοιπόν από την ε, ίδια χώρα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Συνεχίζουμε και δίνω τον λόγο στον συνάδελφο. Ευχαριστώ κύριε Σάκη αγαπητοί προσκεκλημένοι, κύριοι και κυρίες εμπειρογνώμονες, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό εκ μέρους Επιτροπής Ένβη. Έχω την τιμή να προεδρεύω το δεύτερο channel για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό των ε, ενδοκρινικών διαταραχών και πώς μας επηρεάζουν. Έχουμε τρεις ε, επιφανείς επιστήμονες και τοξικολόγους, τον κύριο Μαντοβάνη ε, από το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, τον κύριο Ντάνιελ Δίτριχ και τον κύριο Μάρτιν Όλαν. Και μετά θα κάνουμε την συζήτηση και αρχίζω με τον καθηγητή Μαντοβάνη, τον οποίο δίδω αμέσω το λόγο. Καλήσαμε εσμέρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Είμαι επιστήμων, εργάζομαι στο Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και το θέμα μου είναι ποιες περαιτέρω μελέτες πρέπει να κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να διευθετήσουμε το θέμα τον, του αντικτύπου στην υγεία των ε, ενδοκρινικών διαταραχών. Πώς μπορούμε να προλάβουμε τέτοιου είδους γεγονότα. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι το θέμα αυτό των ε, ενδοκρινικών ε, διαταραχών δεν είναι ένα θέμα το οποίο άρχισε να μας απασχολεί τώρα. Υπάρχουν ε, δεδομένα επιστημονικά τα οποία γνωρίζουμε εδώ και καιρό και η πολιτική που λαμβάνουν τις αποφάσεις, οι επιστήμονες και κυρίως ο κόσμος υποβάλλουν ερωτήματα στην επιστημονική κοινωνία η οποία πρέπει να απαντήσει. Πρώτα απ' όλα, οι διαταράκτες αυτοί είναι διαφορετικοί, πολλαπλοί. Βρίσκονται ακόμη και σε φυσικές ουσίες, σε ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στα τρόφιμα, αλλά στα βιοκτώνα, στα καλλιντικά, στα φυτοφάρμακα, στα ζυζανιοκτώματα. Ε, προκαλούν παρενέργειες, άρα αποτελούν μέρος μελέτης της τοξικολογίας και κάτι το οποίο είναι ιδιάζον είναι ότι το ενδοκρινικό σύστημα είναι πολύπλοκο και είναι αυτό που δίνει στον οργανισμό διάφορα μηνύματα. Τι σημαίνει. Αν λοιπόν αλλοιωθεί κάποια ορμόνη στο σύστημα το ενδοκρινικό, Ε, μας επηρεάζει και μπορεί σε όλα τα στάδια της ζωής να επηρεάσει τον άνθρωπο. Και τα δύο φύλλα συγκεκριμένα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς κατά τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης επηρεάζουν αυτοί οι διαταράκτες τη ζωή του ατόμου αργότερα. Σύμφωνα λοιπόν με τον παρόντα κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τους εντοπίσουμε πρώτα απ' όλα αυτούς τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να ακολουθήσουμε δύο βασικά στάδια. Πρώτα απ' όλα έχουμε ακόμη και στον τομέα της ε, ε, ζωολογίας ε, διάφορες προσεγγίσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Και πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και δεύτερον πώς μπορούμε ε, να ορίσουμε στα διάφορες δοκιμές που γίνονται περισσότερες ε, στόχους για τους ε, ε ενδοκρινικούς διαταράκτες για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την δημόσια υγεία και να την προστατεύσουμε. Okay, excuse me, beg your pardon. So, the problem for non-animal approach. Το πρόβλημα για τις προσεγγίσεις που δεν αφαιρούν το ζωικό βασίλειο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι δράσης, πολυάριθμοι, ε, όλο και περισσότεροι. Είναι όμως και πιο αποτελεσματικοί, όλο και περισσότερα. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλές πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά μας και πρέπει εμείς να τις λάβουμε υπόψη πριν να πάρουμε τις διάφορες αποφάσεις. Αλλά ε, πρέπει να εξετάσουμε ε, μπορούν να προβλέψουν τις παρενέργειες. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη λήψη αποφάσεων ε, όταν ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διάφορες δοκιμές in vivo και τα διάφορα κριτήρια που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και διάφορες ε, θεωρήσεις ε, ποιοτικής ε, αξιολόγησης. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε σε επίπεδο κυταρικό και μοριακό πώς μπορούμε να καταλάβουμε εάν υπάρχει κάποια παρενέργεια από την παρουσία αυτών των διαταρακτών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε εάν μπορούμε να προβλέψουμε αυτές τις ε, παρενέργειες, πώς θα κάνουμε μία νέα αξιολόγηση, ώστε να δούμε πώς με θα μπορέσουμε βάσει κάποιων μηχανισμών να επιλέξουμε ποιοι είναι ποιοτικοί. Δηλαδή, αν υπάρξει κάποια βλάβη στον θηριοειθή αδένα. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε με μία στρατηγική να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις ενδείξεις και τα γεγονότα για να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή λύση. Τα λέγω κάπως βιαστικά όλα αυτά. Ποιες ορμόνες είναι πολύ σημαντικές. Τα εστρογόνα, τα ανδρογόνα και με, για να δώσω ένα παράδειγμα, και Φερρυπίν, εάν έχουμε ξέρουμε ότι ο διαβήτης μπορεί να προκληθεί από την, ε, κάποιους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα θέματα, τα οποία είναι θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, μεταξύ άλλων τον διαβήτη και άλλες ε, ε, μεταβολικές ε, ασθένειες να τις εξετάσουμε λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες, αποδείξεις και Εγώ πρέπει να πω ότι ως Ευρωπαίος πολίτης μπορώ να ε, δεχθώ ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε τους ενδοκρινικούς διαταράκτης, αλλά πρέπει να πω ότι πραγματικά αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να εντείνουμε την έρευνα ώστε να κάνουμε αξιολόγηση του κινδύνου. Είπαμε ότι υπάρχουν διάφοροι επιμολυντές οι οποίοι βρίσκονται μακροπρόθεσμα ε, στο περιβάλλον και μας επηρεάζουν. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε τέτοιου είδους προβλήματα, διότι υπάρχουν προβλήματα με το περιβάλλον, με τα είδη διατροφής και ε, θα επηρεάσουν και τις επόμενες γενιές. Τι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει Να κάνουμε λοιπόν αξιολόγηση του κινδύνου, μείωση του κινδύνου και στρατηγικές ανθεκτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να έχουμε ε, βιολογικούς δείκτες που θα τους προβλέψουμε για να προστατεύσουμε το ζωικό βασίλειο και τον άνθρωπο. Επίσης θα έπρεπε να έχουμε διάφορους ε, ε, ε, ε, τοξικολογικούς ε, αριθμούς αναφοράς αν θέλετε. Επειδή πρόκειται για ένα πολύπλοκο πρόβλημα, δεν θα πρέπει να χαθούμε μέσα σε αυτό. Πρέπει να το αποφύγουμε. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας να τις διασταυρώσουμε, να τις ενσωματώσουμε, να τις εκμεταλλευτούμε, να τις, να τις χρησιμοποιήσουμε και πρέπει πραγματικά να έχουμε μια ειδικά στοχευμένη έρευνα για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα άτομα τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο, τους υπεύθυνους για την διαχείριση ε, κινδύνων, εκτός και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια, διότι ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, και να προσπαθήσουμε να ε, πληρώσουμε τα κενά ενημέρωσης και γνώσεις που υπάρχουν με τη συνδρομή των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Δημόσιας Υγείας και Έρευνας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Και θα συνεχίσουμε αμέσω με τον επόμενο μιλητή από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντζας. So, Okay. So um, I'll start with the title. Synthetic endocrine disruptors at present human exposure are no. Συγγνώμη από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας. Είναι ο καθηγητής Νταν Τίτρης. Εγώ θα τονίσω ότι η, σύνθετα, η συνθετική ενδοκρινική διδράκτη αυτή τη στιγμή δεν αποτελούν κίνδυνο από για την ανθρώπινη υγεία παρά τα όσα ακούσαμε μέχρι τώρα. Να πιστέψουμε στους ορισμούς. Τι είναι η ενδοκρινική διατεράθεση. Έχουμε τη δήλωση του 2013, έχουμε τον ορισμό ΩΣΑ ή του ΠΟΕ, αλλά δεν έχει και σημασία. Ορίζονται οι, οι, αλλά δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα στους συνθετικούς και τους ε, φυσικούς που είναι εξωγενεί σε βάση περιπτώσει σύνθετοι παράγοντες που μπορεί να αλλάξουν, να επηρεάσουν. Αυτό είναι ο ορισμό. Ας πάμε στους φυσικούς. Εκεί έχουμε τη ζάχαρη, γλυκόζη, ζαχαρόζη, φρουκτόζη, ε, ισοφλαβόνες, ε, που παράγεται από την κίτρινη μοστάρδα που καταναλώνεται καθημερινά. Ποια είναι τα αποδεκτά όρια. Τι είναι αποδεκτό κοινωνικο-οικονομικά σε σχέση με την έκθεση, την πραγματική έκθεση. Η ΕΚΑ μίλησε για ελαχιστοποίηση της έκθεση. Η Κομισιόν μίλησε για το βάρος της απόδειξης. Επίσης έγινε λόγος για εντοπισμό του κινδύνου και η ΕΚΑ μίλησε για εντοπισμό κινδύνου, αξιολόγηση κινδύνου και μετά διαχείριση κινδύνου. Μπορείς να διαχειριστείς τον κίνδυνο αν τον έχεις εντοπίσει. Αυτές είναι όμως οι σκέψεις που μπορεί κανείς να σκεφτεί όσο όταν μιλά για κριτήρια αποδοχής. Τι είναι το αποδεκτό. Έχουμε ας πούμε για τους ε, ρήπους ε, όπως τις αλφατοξίνες ε, στα τρόφιμα, όπου το αποδεκτό είναι ένας επιπλέον όγκος σε ένα εκατομμύριο κατοίκων. Αυτό όταν μιλάμε για ε, τα φιστίκια, για τα και, διάφορα άλλα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Τώρα έχουμε ανθρώπινες ασθένειες, νόσους που συνδέονται με την έκθεση στους διαταράχτες. Μιλάμε για στηρότητα, για καρκίνο, για διάφορα σύνδρομα του μεταβολισμού, ε, διάφορες ελληματικές ε, νευρικές και συμπεριφορολογικές αλλαγές και ούτε καθεξής. Και επίσης ε, διαβήτης 1 και 2. Και πάλι ο συνάδελφος Αλβέρτο ήδη μίλησε για διάφορες ε, πορείες και υπάρχουν διάφορες μελέτες ε, μιλάμε για in vitro μελέτες, μιλάμε για αδιποκύτταρα ε, που προχωρούν και προκαλούν καρκίνο στο έντερο. Όλα αυτά από τα, τα βλαστοκύτταρα. Έχουμε όμως και τον δέκτη τον γλυκοκορτικοειδή δέκτη, ο οποίος είναι αυτός που καθορίζει πώς θα επηρεαστεί η ανάπτυξη ενός εμβρίου στη διάρκεια της κοίησης. Okay. Αυτό που σας δείχνω λοιπόν εδώ είναι η κατάσταση σε ένα έμβριο. Έχουμε λοιπόν έγκυο τη γυναίκα, παίρνει φάρμακα, ε, γίνεται κάποια αγωγή δηλαδή, ε, ε, ίσως είναι άρρωστη, άρα χρειάζεται κάποια φάρμακα, Έρχεται τη διατροφή που επίσης επηρεάζει το έμβριο, γενετικά στοιχεία και περιβάλλον. Και όταν μιλάμε για περιβάλλον, μιλάμε για αυτούς τους ε, ενδοκρινικούς διαταράχτες. Πώς λοιπόν αυτοί επηρεάζουν το έμβριο. Τώρα αυτό που έχω να σας πω, να σας δείξω, είναι κάπως περίπλοκο αλλά τη ουσία ποια είναι. Πάνω βλέπετε ένα είδος κορτικοειδούς ε, ε, ε, αγωνιστές, εν πάση περιπτώσει, ότι θέλετε να τους πείτε, που πηγαίνουν στην δέκτη και μπορεί να οδηγήσουν σε αντιπογέννηση. Μετά έχουμε τους ανταγωνιστές που εμποδίζουν, μπλοκάρουν αυτή τη δράση. Βλέπουμε λοιπόν μια γυναίκα η οποία εκτίθεται σε έναν μεγάλο αριθμό φαρμάκων, μάλλον σε, φάρμακα για τη θεραπεία κάποιας ε, ασθένειας και αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ο συνδυασμός in silico, in vitro και in vivo πειραμάτων που μπορούν να προβλέψουν ποιος είναι ο θεραπευτικός δείκτης, δηλαδή πού ε, βρίσκεται το όριο μεταξύ της θεραπείας της μητέρας και της έκθεσης του ε, εμβρίου. Και αυτό που βλέπουμε εδώ είναι το περιθώριο έκθεσης, δηλαδή ασφάλεια ανάμεσα στην πραγματική έκθεση της μητέρας και του τι λαμβάνει τελικά το έμβριο. Και εδώ φτάνουμε γύρω στα 300 και 10.000 ε, άτομα. ντάιτζεν, γενιστέν και Δυσφενόλη. Πόσο δυνατέ είναι αυτοί οι αγωνιστές που είπαμε, οι δραστικές ουσίες, ας τις πούμε έτσι. Ποια είναι η δόση δηλαδή η οριακή. Το... Αυτές οι ουσίες ε, ε, ρυθμίζουν τον, ε, την υποδοχή από τον στεροειδή. Θα δούμε κατά πόσο θα επηρεαστεί το, σε ποιο επίπεδο και μετά επηρεάζεται το έμβριο, ώστε να αναπτύξει αργότερα διαβήτη τύπου 2. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να δούμε ποια είναι η κατάσταση της γυναίκας στη διάρκεια της σκήσης. Και εδώ τα πράγματα αλλάζουν α, σε τεράστιο βαθμό. Πρόσφατα στοιχεία έχουμε από την... υπηρεσία Food and Drug των ΙΠΑ που εξέτασαν αυτή την ε, κατάσταση. Τα διάφορα ιστρογόνα έχουν αυξηθεί κατά 10 9 Ε, μονάδες, ενώ ταυτάχρονα, αν δούμε Dadsen ε, και Τζένιστεν αυτά κατεβαίνουν ε, κατά 10 με 100 φορές. Ενώ η δυσφενόλη α είναι 100.000 φορές χαμηλότερη. Οπότε το ερώτημα είναι, όταν ε, ένας, ε, ε, είναι κατά πόσο αυτός ο παράγοντας δυσφενόλης α μπορεί να επηρεάσει στη διάρκεια της ευκαιμοσύνης, στη διάρκεια της σκήσης, θα έπρεπε να είναι το ίδιο δραστήρια όπως και τα ενδογενή συστήματα. Δεν είναι όμως, άρα λοιπόν είναι το θέμα πόσο μεγάλο είναι ο κίνδυνος ή όχι άλλο που θέλουμε να σε δείξουμε είναι η βυσφενόλη F. Εδώ έχουμε μια έκθεση που κάναμε εμείς στο δικό μας εργαστήριο και έχουμε συγκρίνει τη δυσφενόλη Α και τη δυσφενόλη F από την κίτρινη μοστάρδα. Η F είναι πολύ πιο ψηλή η παρουσία της στην έγκυο γυναίκα από ότι η Α. Το θέμα είναι λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ένας κανονισμός ε, της δυσφενόλη ε, α σε σύγκριση με τη ζάχαρη και τη δυσφενόλη F. Επανέλθουμε στον Μπερνάρ που είπε, είπατε ότι πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση, αλλά θα πρέπει να γίνει για όλους τους ρήπους και όλα, όλα τα, όλες τις ουσίες και τη ζάχαρη μεταξύ αυτών. Έχουμε και μια μελέτη που εξετάζει την κατάσταση για το πώς η δυσφενόλη α επηρεάζει τις ε, άλλες διάφορες ουσίες και δεν υπάρχουν ε, πορίσματα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις που να είναι μετρήσιμες. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια συγκεκριμένη δόση. Το θέμα είναι υπάρχει πραγματικά πρόβλημα με τη δυσφυνόλη α, αν και μας ανησυχεί πολύ αυτή η ουσία για κάποιους κατανόητου λόγους. Επόμενο παράδειγμα, όπου επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νομίζω την κοινή λογική, είναι η κατάσταση με την DDE. ότι έχει μεγάλη επιρροή στην παχυσαρκία και στο διαβήτη. Βλέπουμε όμως ότι μειώνεται η συγκέντρωση DDE στην γενικό ευρωπαϊκό πληθυσμό και τα στοιχεία που σας δείχνω δεν, δεν είναι πρόσφατα, είναι του 2000, είναι στοιχεία 18 ετών και ήδη είμαστε πάρα πολύ χαμηλά. Εδώ έχουμε δεκαετή στοιχεία για την παχυσαρκία από τον ΩΣΑ. Πού έχουμε παχυσαρκία και πού συνεχίζεται η χρήση του DDTDDE. Βλέπουμε Ινδία, Κίνα, Ινδονησία μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσαν ε, σε μεγάλες συγκεντρώσεις το DDE, αλλά δεν επικρατεί η παχυσαρχία. Όμως παχυσαρχία υπάρχει σε όλες τις χώρες που έχουν απαγορεύσει το DDE, εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Πάλι είναι θέμα κοινή λογική. Οι χαμηλότερε συγκεντρώσει ξαφνικά οδηγούν σε μεγαλύτερη ανταπόκριση. Αυτό είναι αντίστοιχο, αντίθετο συγγνώμη, με την επιστημονική αντίληψη. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια με, με, με τα ενδοκρινικά χημικά Όμω, ποιο είναι το θέμα και είπα ανέφερε τη ζάχαρη από νωρί. Βλέπουμε την κρίση της ε, ζάχαρης ε, στις ΕΠΑ ε, και την παχυσαρκία του πληθυσμού. Βλέπετε ότι η παχυσαρκία συμπίπτει με την μεγάλη πρόσληψη ζάχαρης, ενώ αν δείτε κάτω αριστερά πώς αυξήθηκαν οι αλυσίδες fast food, και πώς η ε, υπερβολική πρόσληψη λίπους και ζάχαρης ελαίων ε, ταυτόχρονα έχουν οδηγήσει στην παχυσαρκία. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα όσον αφορά την παχυσαρκία, την ε, αύξηση λίπους και τον διαβήτη τύπου 2. Όχι, λοιπόν, Το okay. είναι. πολύ ποσά. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι βάσιμα τα στοιχεία περί των, δημο... των ενδοκρινικών Τουλάχιστον όχι με βάση τα επιστημονικά πορίσματα. Λυπούμε που το λέω αυτό, αλλά έτσι είναι. Τώρα, Ε, εμείς έχουμε δει ότι η έκθεση στους ενδοκρινικούς διαταράχτες είναι πολύ χαμηλή για να επηρεάσει το παιδί. Ε, έκθεση ωστόσο στην ζάχαρη σίγουρα θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην υγεία, καθώς και η υπερβολική κατανάλωση λίπους και θερμίδων ε, θα έχει ε, αντίθετο αποτέλεσμα, αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν υπάρχουν ε, και είναι τεκμηριωμένα. Σε σχέση λοιπόν με τα μέτρια αυτά τις μέτρες επιρροές του των, των ενδοκρινικών αδιατρακτών στην υγεία και μάλιστα έρχομαι από πρόσφατο συνέδριο ενδοκρινολόγων, ε, το ερωτηματικό παραμένει με την εξαίρεση φυσικών ε, συνόλων όπως οι ισοφλαβόνες, η ζάχαρη σημαντικές ασθένειες, ε, ε, διαβήτης 2, είναι αδύνατον να συνδεθεί ως αίτιο ε, με τις, τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Γιατί είναι πολύ χαμηλές οι συγκεντρώσεις που βρίσκουμε στα άτομα που εκτίθεται. Θα πρέπει λοιπόν να καλύπτεται η αιτιότητα και όχι η πιθανότητα Είδα τις διαφάνειες της ε, πρότασης Κομισιόν και με χαρά διαπίστωσα ότι το λαμβάνουν αυτό υπόψη. Ε, θα πρέπει να δούμε in vitro και in vivo ε, τεστ που έχουν γίνει. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πραγματική ανθρώπινη έκθεση, δηλαδή ο κίνδυνος. Θα πρέπει να εξετάσουμε πιο πιθανές εξηγήσεις στις ε, για ανθρώπινες ασθένειες ε, πριν να αναφερθούμε στη σύνδεση με τους ενδοκρινικούς διαταράκτε. Με αυτό κλείνω και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Well then, thank you, professor. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Να ρωτήσω τώρα τους συνεργάτες μας αν είναι έτοιμη η βιντεοδιάσκεψη. Σχεδιασμός στο Λονδίνο και σας δίνω το λόγο. Αξιότιμη πρόεδρε, Αξιότιμοι συνάδελφοι, επιστήμονες, ευχαριστώ που μας δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σήμερα για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Τι ξέρουμε λοιπόν για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες είναι το σύστημα επικοινωνίας του οργανισμού για τις ε, ε, κατάλληλες ανταποκρίσεις περιβαλλοντικές συνθήκες. Συνήθως είναι μεταβατικές αυτές οι ανταποκρίσεις και ο λόγος του ενδοκρινικού συστήματος είναι να διατηρεί την ομοιόσταση, δηλαδή να επαναφέρει το status quo όταν επανέλθουν οι συνθήκες στο κανονικό, όπως το ενδοκρινικό σύστημα, όμως έτσι και ο ρόλος ε, του ενδοκρινικού συστήματο στην ε, ε, στα πρώτα τη ζωή είναι να ορίσει τον κανόνα, το, το status quo αυτό, με βάση τις ε, ε, κρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες. Συγγνώμη, παρακαλώ, πιο σιγά να μιλάτε παρακαλώ, γιατί δεν μπορείς να σας παρακολουθήσουν οι διερμηνείς. Λίγο πιο αργά να μιλάτε, να διαβάζετε κλασική άποψη λοιπόν του ενδοκρινικού συστήματος είναι ότι πρόκειται για μια σειρά από αδένες που επικοινωνούν μεταξύ τους ε, εκρήγνοντας ε, χημικούς διαβιβαστές στους οποίους μεταφέρει το αίμα, ε, τις ορμόνες συγκεκριμένα. Όμως ε, το ενδοκρινέ σύστημα τελικά συνειδητοποίησαμε ότι περιλαμβάνει και άλλα όργανα όπως ε, είναι το πάγκρες και άλλα χημικά σήματα μεταξύ και εντός και που δεν έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία του αίματος. Ε, τελικά το ενδοκρινέ σύστημα επηρεάζει κάθε όργανο και κάθε κύτταρο του σώματος. Ε, γιατί πρέπει να μας ανησυχεί η ενδοκρινική διαταραχή. Η ε, ενδοκρινική διαταραχή σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα αυτό επικοινωνίας. Και υπάρχουν πιστικά, πιστικές ότι πραγματικά κάτι πάει άσχημα, κάτι πάει στραβά. Ε, υπάρχουν περισσότερες νόσοι που σχετίζονται με ε, την λειτουργία των ορμονών όπως η νορμονική καρκίνη, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού προστάτη των όχεων, ε, η πρόψιμη, η πρόορη μάλλον εφηβεία, η κρυψορχία, αταραχές στη σύλληψη, μείωση του αριθμού σπερματοζωαρίων, μεταβολικές ασθένειες όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. μεταξύ των 15 έως ε, είναι ο πιο συχνός, το πιο συχνό κακό ήθες νεόπλασμα ε, στον άντρα, ακριβώς η καρκίνη στις γονάδες, ε, στους όρχες. Και δείχνουν τα στοιχεία επίσης για τον καρκίνο του μαστού ότι οι χώρε με το χαμηλό εισόδημα αρχίζουν να φτάνουν τα ποσοστά των χωρών με το υψηλό εισόδημα και οι ορμόνε σχετίζονται με νοσήματα που έχουν να κάνουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου, όπως είναι αυτισμός ή ή διαταρχές ελληματικής προσοχής, μείωση του IQ. Η αύξηση των ε, τάσεων αυτών ε, δείχνει ότι η γενετική, παραδοσιακή γενετική παράδοση από μόνοι τους δεν μπορεί να εξηγήσουν αυτές τις τάσεις. Ε, μελετώντας μεταναστευτικούς πληθυσμούς που πηγαίνουν από το μία χώρα στην άλλη, βλέπουμε ότι η πρώτη γενιά δεν αποκτάει τον ίδιο κίνδυνο να αναπτύξει ένα νόσημα στη χώρα υποδοχή, αλλά η δεύτερη ναι. Και αυτό δείχνει ότι το περιβάλλον, τρόπο ζωής επηρεάζουν τη δημιουργία νοσημάτων. Δεν μπορεί η αύξηση να εξηγηθεί μόνο απλά με τις αλλαγές στο screening, τις διαγνώσεις ή τη γέρανση του πληθυσμού. Με βάση μάλιστα την τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, <clears throat> το βάρος νόσων από περιβαλλοντικό κίνδυνο παραμένει παράλλακτο από το 2002 και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσετε κανεί παρασιτικές, διατροφικές ε, και μεταδοτικές νόσοι, αλλά δυστυχώς αυτό αντισταθμίστηκε και από την άψη μη μεταδοτικών ασθενειών. Δεν ε, είναι εύκολο να λυθεί το πρόβλημα. Πολλές είναι χρόνιες παθήσεις που απαιτούν διαρκή θεραπευτική αντιμετώπιση. Και αυτό επιβαρύνει τα ασφαλιστικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Η υγεία στα πρώτα χρόνια της ζωής ε, καθορίζει τη μελλοντική υγεία του ενηλίκου. Ο Βρετανός επιδημιολόγος David Barker είναι αυτός που μίλησε για αυτήν την υπόθεση μέσα του 80. Παρακολούθησε το γεγονός ότι από τι ελλείψει τροφίμων στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι γυναίκες, οι έγκυε, οι οποίε πραγματικά λιμοκτονούσαν, γέννησαν παιδιά που αργότερα ανέπτυξαν ε, ε, κίνδυνο, είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν μεταβολικές καρδιαγκιακέ παθήσεις. Η επιγενετική είναι μια πολύ σημαντική επιστημονική εξέλιξη των τελευταίων 10-15 ετών και δεν μας εκπλήσει το γεγονό ότι οι ορμόνες παίζουν σημαντικό ρόλο για τις επιγενετικές αυτές τροποποιήσεις που μπορεί να μεταφερθούν μερικές από τις επόμενες γενιές, ακόμη και αν δεν έχουν εκτεθεί. Έχουμε τη διεθυλστιλβιστρόλη, ένα ισχυρό ιστρογόνο που αποδεικνύει αυτή την έννοια. Οι γυναίκες που έπαιρναν αυτό το φάρμακο ε, στην αρχή της κοίησης ε, αντιμετώπισαν ε, προβλήματα και οι γυναίκες τους είχαν αυξη... οι κόρες τους συγγνώμη, είχαν αυξημένο <laughs> κίνδυνο καρκίνο του μαστού, προβλήματα γονιμότητας και άλλα γυναικολογικά ζητήματα, οι δε γη τους, προβλήματα αερογεννητικής φύσεως ε, και ενδεχόμενο ανάπτυξη καρκίνου των όρχεων. Και βέβαια κίνδυνο ακόμα μεγαλύτερο για τα εγγόνια. Υπάρχει μια κακή προσαρμογή στο περιβάλλον από ό,τι φαίνεται η έκθεση σε παρόντες κινδύνου είναι κάτι που θα το δούμε δεκάδες ε, χρόνια ε, και για τις επόμενες γενιές θα είναι ε, κάτι που θα αντιμετωπίσουν ως πρόβλημα. Είναι πολύ παραγωγικές συνώσεις, δεν υπάρχει μια αιτία, πολύ περιβαλλοντικοί παράγοντες αλληλένδετοι που έχουν να κάνουν και με τη διατροφή, την καθιστική ζωή, το άγχος, της χημικές ουσίες. Και δεν θα πρέπει αν έχουμε στοιχεία που υποστηρίζουν το ρόλο ενό παράγοντα, να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο παράγοντα που επίση επηρεάζει. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι ο ρόλο των χημικών ουσιών. Μπορεί ε, τα χημικά να διαταράξουν το ορμανικό σύστημα. Ναι, και το γνωρίζουμε εδώ και δεκαετία, ε, μην πω έναν αιώνα, για τα συνθετικά χημικά. Ε, χαμηλές τρογονικές ιδιότητες της φυσενόλης α ανακαλύφθηκαν το 1930 όταν ψάχναμε συνθετικά χημικά για να αντικαταστήσουν το φυσικό ιστρογόνο που είναι ακριβό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την σεξουαλική ικανότητα των ανδρών, 80 και 90 έγιναν μελέτε in vitro και μελετήθηκαν πολλά χημικά που μπορούν να μιμηθούν τα ιστρογόνα, όπω κάποια ζυμοκύτταρα ή ε, διατηρημένα ε, καρκινικά κύτταρα του μαστού. Και είδαμε ότι έχουν και αυτά δράση παρότι μικρότερα από τα φυσικά ιστρογόνα, φυσικές ορμόνες. Συνάδελφος ε, Σίλβα και ο καθηγητής Κόρτεν Κάμπ δημοσίευσαν ε, ένα έγγραφο, Something from Nothing λέγεται, με βάση κάποια στοιχεία από ζυμοκύτταρα ε, χρησιμοποίησαν ένα μείγμα έξι χημικών σε συγκεντρώσεις που δεν θα είχαν ανιχνεύσιμες επιπτώσεις αλλά ως μείγμα είχαν τα, τα χημικά αυτά επίπτωση Τι γίνεται λοιπόν, πώς επηρεάζουν αυτά την υγεία το περιβάλλον. Επίσης, Μπορεί να μην είναι τα ίδια τα αποτελέσματα στι διάφορε μελέτε. Σίγουρα είναι ε, να κλειδί κατά κάποιο τρόπο οι ορμόνε για έναν υποδοχέα ε, που είναι κλειδαριά, αλλά υπάρχουν διαφορετικοί υπότυποι υποδοχέων μπορεί να βρίσκονται στο πυρήνα και στην επιφάνεια, στο κοιτόπλισμα ή σε κυταρικά οργανίδια. Ο καθηγητής Angel Νατάλ βρήκε ότι η σε κυταρικα οργανιδια ο καθηγητή angel Natal βρηκε οτι η δυσφενολη α είναι το ίδιο ισχυρή με το φυσικό ιστρογόνο για την απελευθέρωση ινσουλίνης από τα παγκρατικά κύτταρα β ή τα νησίδια του Λάγκερχανς και θα πρέπει να μελετάμε ε, και να λαμβάνουμε ε, επιφυλακτικά υπόψη μας τα αποτελέσματα μελετών που μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους. Τι στοιχεία έχουμε για τα χημικά. Υπάρχουν επαρκή επιδημιολογικά στοιχεία ε, για το ρόλο των χημικών. Παραδείγματο χάρη, μία σχέση μεταξύ τη έκθεση στα ζενεκτώνα και του καρκίνου του προστάτη. Σε μεταναλύσει αποδείχθηκε αυτό. Και έγιναν και διάφορε μελέτε που δείχνουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τη έκθεση γυναικών σε φταλικέ ενώσει ε, και την ε, προκτογεννητική απόσταση στα αγόρια, <clears throat> που είναι μειωμένη. Και αυτό δημιουργεί γενετικά προβλήματα. Αυτό περιπέκεται από το γεγονό ότι οι άνθρωποι περιβάλλον εκτίθεται ταυτόχρονα αλλά και κατακολουθία σε διάφορα χημικά και τα διάφορα μοτίβα έκθεσης ε, είναι πιο πολύπλοκα. Παραγωγή κατανάλωση για μηχανικών χημικών αυξάνεται. Η χρήση του σε προϊόντα και διάφορα άλλα είδη ποικίλει. Άρα δεν μιλάμε για υψηλή δόση και οξία έκθεση, αλλά σε χρονικά επίπεδα έκθεσης χαμηλά. Σε και σε πολλαπλές χημικές ουσίες. Υπάρχει πολλαπλή αιτιότητα. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται έρευνα δεκαετιών για να συλλεγούν στοιχεία που θα αποδεικνύουν ή τόσο θα προσπαθήσουν να αποδείξουν, να ψωτικοποιήσουν τον αντίκτυπο της έκθεσης σε κάποιες ουσίες στη Μήτρ. Δεν το έχει πετύχει η ρύθμιση ε, μέχρι τώρα. Πολλές φορές κάνουμε πειράματα σε νεαρά υγιή ζώα υπό ελεγχόμενες και ευέλτιστες συνθήκες ε, για να κάνουμε την παραβολή των ε, αποτελεσμάτων. Τώρα, τα σημερινά τέστα μπορούν να ε, ανοιχνεύσουν ε, την ενδοκρινική διαταραχή. Έξι έχουν ανακαλυφθεί πρόσφατα. Τρεις όμως μέσω ρυθμιστικών ε, δοκιμών. Οι πέντε από τους ερευνητές. και δεν είναι κατάλληλος αυτός, ε, αυτές, ο κύκλος δοκιμών για την ταυτοποίηση δοκρινικών ε, διαταρακτών. Υπήρξε κάποια πρόοδος όπως ε, μετά από την επικύρωση δοκιμών από τον ΟΣΑ, αλλά υπάρχουν κάποια τυφλά σημεία, πρέπει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά. Πέρυσι έγινε ένα εργαστήριο για τη θεωρητική διαταραχή. Μεταξύ άλλων ήταν και ο καθηγητή Μαντοβάνη εκεί. Και συμπέρασμα ήταν ότι η ανείχνευση των θερεδοδικών ε, διατακτών μπορεί να παρακολουθεί λόγω του ότι δεν είναι ικανοποιητικέ οι δοκιμέ στο πλαίσιο του ΩΣΑ. Με τι δοκιμέ μπορούμε να ανοιχνεύσουμε ορισμένου, αλλά όχι όλου του ενδοκρινικού διατάρακτε σήμερα. Ούτε μπορούμε να προβλέψουμε αποτελεσματικά τι επίπτωση θα έχουν στην υγεία το περιβάλλον. Θα πρέπει επίση να δούμε πώ επηρεάζουν τα μείγματα ή πώ μπορεί οι μικρέ δόσει να επηρεάζουν. Αλλά παρόλα αυτά <clears throat> δεν πρέπει να υπεραπλουστεύσουμε τα θέματα αυτά γιατί είναι πάρα πολύ πολύπλοκα. Ολοκληρώνοντα. Τα χημικά δεν είναι ο μόνο ε, παράγοντα από τι ανισχυτικέ τάσει για τι μη μεταδοτικέ ασθένειε, είναι όμως ε, ένας ε, παράγοντα που επηρεάζει. Δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι αποτελεσματικέ παρεμβάσει στον τομέα τη δημόσια υγεία για αλλαγή τη προσωπική συμπεριφορά που έχει να κάνει με τι διατροφικέ συνήθειε, τη φυσική, τη σωματική δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν, μάλλον υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι επηρεάζουν οι αλλαγές στη διατροφή, όπως πρέπει χάρη λιγότερη πρόσληψη ζάχαρης. Αλλά ε, περιμένουμε την πολιτική να πάρει και αυτή τα μέτρα της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αρχίζουμε τώρα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου Ο κύριος Χουίτεμαρ βλέπω πρώτα απ' όλα να ζητά το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι μέλος της ΕΝΒ και της αλλά θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Βλέπουμε επιστήμονες, ακούμε διαφορετικές ιστορίες. Ε, υπάρχει λοιπόν ένας κοινό παρανομαστής μεταξύ όλων αυτών που είπατε, αλλά υπάρχουν και διαφοροποιήσεις, δεν είναι έτσι. Αυτό διαπίστωσα κι εγώ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους παρεμβαίνοντες για την ποιότητα των παρεμβάσεων τους και για το πόσο ε, μετριοπαθώς εξέθεσαν ε, τις επιστημονικές τους παρατηρήσεις. Είδα λοιπόν με πόση προσοχή οι, οι ειδικοί αυτοί οι επιστήμονες αναλύουν την κατάσταση και διαρωτώ με πραγματικά σε σχέση με τις θέσεις της Επιτροπής έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μετριοπάθεια επαναλαμβάνω εκ μέρου των επιστημόνων γιατί είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το θέμα. Πολλές φορές όμως υπάρχει και η βεβαιότητα και εμεί βρισκόμαστε μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων. Βεβαιότητα, βεβαιότητα, μετριοπάθεια, ακούγοντας τι λένε οι επιστήμονες και ακούγοντας και τι έχουν πει στις ε, γνωμοδοτήσεις τους οι εκπρόσωποι της Επιτροπής. Πρέπει να είμαστε όλοι σίγουροι ότι ενεργούμε βάσει της ε, αρχής ε, της προφύλαξης, προειδοποίησης και έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα δημόσιας υγείας που αφορά όλα αυτά τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών και άλλων. Ε, η γεωργία παράγει τα είδη διατροφής που καταναλώνουμε. Αλλά κάποια προϊόντα που χρησιμοποιούμε, κάποιες ουσίες, ε, ακούμε και διαπιστώνουμε ότι είναι επικίνδυνες, άρα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε. Βλέπουμε λοιπόν πόσο στενά συνδεδεμένα και εγκάρσια συνδεδεμένα είναι η, η υγεία του καθενός μας και τα είδη διατροφής που παράγει η γεωργία μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και τι είδους κοινωνία θέλω να έχουμε. Σήμερα βλέπουμε ότι το μέλλον της γεωργίας περνάει από την ε, τα συστήματα ελευθέρων ε, συναλλαγών από μεγάλες εταιρείες. Βλέπουμε ποια είναι τα μοντέλα που ακολουθούνται σήμερα. Βλέπουμε τα μεταποιημένα είδη διατροφής τι, κακό μπορούν να μας κάνουν. Η ζάχαρη φερινής, ε, η υγεία του καθενός, η παχυζαρκία που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα έχουν άμεση σχέση με αυτά που ακούμε. Θα Πρέπει λοιπόν ακούγοντας τι έχουν να πούν οι επιστήμονες να διαπιστώσουμε ότι θα πρέπει όλα αυτά οι πολιτικοί και αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις να το λάβουν υπόψη και να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες στην πολιτική μας. Η υγεία των συνανθρώπων μας δεν πρέπει να είναι η απόλυτη ε, προτεραιότητα ή θα πρέπει να είναι τα οικονομικά αποτελέσματα αυτά τα οποία θα μας ε, καθοδηγήσουν τις αποφάσεις μας. Θα πρέπει να ασχοληθούμε ενδελεχώς με το θέμα για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε αυτό το θέμα. Και πραγματικά αυτή η προβληματική πρέπει να μας απασχολήσει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινέστατα, διότι με τα παρατηρήσεις που κάνατε, με τις παρεμβάσεις σας, με τις επιστημονικά αποδεδειγμένες παρεμβάσεις σας, μας κάνετε να σκεφτούμε πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για όλους μας. Ευχαριστώ. Φοβούμαι ότι ως βιολόγος ε, μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα. Αυτή είναι η βάση της επιστήμης, ότι ακριβώς μπορεί κανείς να αναπτύξει μια υπόθεση και η υπόθεση αυτή πρέπει να αμφισβητηθεί και να αποδειχτεί. Αυτό θα πει η επιστήμη. Διαφορετικά είναι ε, απάντηση στις ερωτήσεις σας θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Η κυρία Εύη είναι η επόμενη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ σας αναφέρω το νέο ότι στην περιοχή του Βένετο, μάλιστα χθες ε, κηρύχθηκε επίγουσα κατάσταση ανάγκης λόγω της ρήπανσης. Είναι ένα ε, σήμα μεγάλης ανησυχίας που προέρχεται από τις περιφέρειες, τους πολίτες και επιβεβαιώνεται και από την δράση του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο προσπαθεί να να ε, προσπαθήσει μαζί με την Κομισιόν να αυξήσει όσο γίνεται περισσότερο την υγεία των πολιτών ε, σε σχέση με αυτήν ε, την σημερινή υπόθεση, δηλαδή τους ενδοκρινικούς διαταράχτες. Πρόκειται φυσικά για ένα εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα με πολλές πτυχές που είναι πολύ δύσκολο να το πλαισιώσουμε και να το περιχαρακώσουμε. Εγώ συνδέομαι με όσα είπαν οι περιπτώσει συνάδελφοι, ότι δηλαδή η ρήπανση του περιβάλλοντος, του αέρα, του νερού, των τροφίμων, των όσων χρησιμοποιούμε καθημερινά, στην ουσία δημιουργούν ένα ναρκοπαίδιο. Δημιουργεί η ρήπανση ένα ναρκοπαίδιο και μέχρι σήμερα ε, πιστεύαμε ότι είμαστε βέβαιοι, ενώ όταν διαπιστώσουμε πόσο περισσότεροι κίνδυνοι μπορεί να κρύβονται, ε, κανείς τα χάνει και, και μπορεί να κρύβονται κίνδυνοι για τις μελλοντικέ γενιές και αυτό είναι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, ε με ε, περισσότερο, οι επόμενες γενιές. Εγώ θέλω να αναφερθώ στο ρόλο της επιστήμης. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό το μεγάλο ζήτημα. Θέλω να ρωτήσω αυτούς, όλους τους εμπειρογνώμονες που είναι σήμερα εδώ σε σχέση με το ποιος θα πρέπει να είναι ο δημόσιος ρόλος στην επιστημονική έρευνα. Γιατί πολύ συχνά είδαμε ότι η παρέμβαση από πλευράς ε, ιδιωτικών συμφερόντων μπορεί σε κάποιο βαθμό να προσανατολίσει και να καθορίσει τις πολιτικές επιλογές και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω από τους εμπειρογνώμονες δεν θεωρείτε ότι ο ρόλος της δημόσιας έρευνας θα έπρεπε να είναι ε, όλο ένα και πιο υποστηριζόμενος ε, για να μπορέσει να πετύχει οποιοδήποτε είδος απόφασης να βασίζεται αποκλειστικώς στην επιστημονική έρευνα, στην ε, εξένταση την ε, επανεξέταση των, από πλευράς των ομολόγων, δηλαδή συμμετοχή ολόκληρης της επιστημονικής κοινότητας με τρόπο ώστε να μην μένουν σημεία ε, σκιασμένα ή να μην υπάρχει αδιαφάνεια. Και η τελευταία ερώτηση αφορά το project που ανέφερε ο καθηγητής Ματοβάνη, που από το, χρηματοδοτήθηκε από το Horizon 2020 και θα ήθελα να έχω περισσότερες πληροφορίες, να δούμε δηλαδή πώς ακριβώς έγινε, γιατί πιστεύω πως ακριβως γινεται γιατι πιστευω πως υπαρχει μια καλή πρόταση. Είναι καλό το project και θα ήθελα να έχω περισσότερες ε, πληροφορίες. Μήπως θα έπρεπε να δούμε λοιπόν ότι είναι ένα αξιόλογο πρόγραμμα γιατί έτσι δεν χρησιμοποιείται εκεί, δεν χρησιμοποιούνται ούτε ε, και τα ζώα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις των ε, ομιλητών μας που είναι πανεπιστημιακοί. Πραγματικά ε, και εγώ σύμφωνα με αυτή την ερώτηση. Η κυρία Ροζιέ. Σας ευχαριστώ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και αποκαλύπτεται από αυτά που είπαν οι επιστήμονες πόσο πολύπλοκο είναι το όλο θέμα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πραγματικά πώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί. Ήταν ε, εξαιρετικά διαφωτιστική τελευταία παρέμβαση. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά το μηχανισμό και βλέπουμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις ε, που οφείλονται. Βεβαίως θα πρέπει να, γίνουν να υπάρξει περισσότερη χρηματοδότηση της δημόσιας έρευνας για να έχουμε όλο και περισσότερο εμπεριστατωμένες γνώσεις. Εμείς όμως δεν είμαστε ερευνητέ, δεν είμαστε επιστήμονες αν θέλετε στον τομέα αυτό. Καθένα επιστήμονε στον τομέα, το λέω όχι εδώ. Και Ξέρουμε ότι οι αποχρώσεις διαφορές είναι πολύ σημαντικές και όλο περισσότερε γνώσει έχουμε τόσο καλύτερα, αλλά εμείς δεν έχουμε το μέτρο στη διαθεσή μα. Ξέρουμε ότι η βιομηχανία έχει δικές της ε, επιλογές ανάλογα με το τι προϊόντα παράγει και σε ποιον απευθύνεται. Και βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις διαφορές στην έρευνα ε, και είναι πολύπλοκο το θέμα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ξέρουμε ποιες είναι οι σαφείς γραμμές που μπορούμε να ακολουθήσουμε ε, για να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχή της προφύλαξης εμείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον καθορισμό των κριτηρίων μιλάει για αυτή την αρχή της προφύλαξης και κυρίως τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Αλλά εμβαθύνοντας όλο και περισσότερο, διότι η έρευνα και η... μας βοηθάει πάρα πολύ. Ας μην προσπαθήσουμε όμως να ανατρέψουμε το μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Βεβαίως πρέπει να έχουμε γνώσεις, αλλά υπάρχουν αρχές τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε και ιεραρχώντας τις ε, προτεραιότητές μας, πρέπει να πω ότι πρωταρχικό μας μέλημα είναι η υγεία των πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Βλέπω ότι θέλουν να απαντήσουν οι επιστήμονες που έχουμε καλέσει. Κύριε Μαντοβάν. Thank you. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες. Οι ερωτήσεις αντικατοπτρίζουν ε, τις προφανείς και λογικές αμφιβολίες αντικατοπτρίζουν τον προβληματισμό και των ίδιων ε, των επιστημόνων. Γιατί όλοι μας ε, μελετούμε διαφορετικές επιτυχίες. Εν μέρη είναι αλήθεια και εν μέρη όχι. Η επιστήμη ζει από τη συζήτηση. Δεν μπορεί όμως να συνεχίσει να ζει με ατελείωτες συζητήσεις. Εάν κάνεις ρυθμιστική επιστήμη, δηλαδή μετάφραση της έρευνας σε επιστημονική στήριξη για αποφάσεις, εκεί για λήψη αποφάσεων, εκεί κάπου πρέπει να καταλήξει. Να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, πορίσματα. Και αυτό βέβαια μετά από συνένεση. Ε, ε, μετά από μελέτη όλων των συμβολών. Αυτή τη στιγμή επικρατεί γενική συνένεση ότι οι διαταράχτες είναι ζήτημα αυτό κάθε αυτό. Ε, πρέπει να, όμως να ε, οριστεί, να εντοπιστεί. Ε, τώρα, η ευρωπαϊκή πολιτική λαμβάνει αποφάσεις καταρχάς για την αναγνώριση και τον εντοπισμό αυτών των χημικών ουσιών. Αλλά όπως προσπάθησα να εξηγήσω στην δική μου παρέμβαση και μιλώ για τον εαυτό μου και μόνο εξ μου, η αξιολόγηση κινδύνων σε πολλές πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να ξεπεραστεί ο στάδιο, να αποφευχθεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πόσο πολύ θα πρέπει να περιορίσουμε, <coughs> δηλαδή σε ποιο βαθμό θα πρέπει να προστατεύει ο νόμος για τις ε, διαρκείες εκθέσεις, αν υπάρχουν τέτοιες, ε, διαρκείες εκθέσεις, εφόσον και είναι και διαρκείες ο κίνδυνος. Εγώ δεν είμαι επιδεμιολόγος και δεν ήθελα να απαντήσω σε αυτό το θέμα. Η απάντησή μου, ωστόσο, ακούγοντας τις περισσότερες σας τους άλλους πιο εμπειρογνώμονες που έχουν κάνει επιδημιολογικές μελέτες, η απάντηση είναι ότι ίσως και να έχουμε πρόβλημα, για να το πω έτσι πιο μετριοπαθώς, τουλάχιστον για τους αναπτυσσόμενους οργανισμούς. Και ξέρω ότι ο Ντάνιελ ε, θα, θα απαντήσει πιο έντονα. Δεύτερο θέμα, δεύτερη αντίδραση είναι... Ρυθμιστικές λοιπόν σχέσεις ε, με την επιστήμη. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα τονίζει ότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκού επίπεδου έρευνα, από το Horizon 2020 ας πούμε, ε, θα πρέπει να χρηματοδοτεί τέτοιου είδου έρευνα. Έρευνα νομοθετικού τύπου για τη βιομηχανική ασφάλεια, για την εργασιακή ασφάλεια, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τους εργαζόμενους και ε, περιβαλλοντική ασφάλεια. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και όχι μόνο οι ενδοκρινικές διαταράκτες φυσικά. Να είναι σφαιρική η ευρωπαϊκή έρευνα και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε πιο πολύ έρευνα που χρηματοδοτείται από τα δημόσια κονδύλια και άρα περισσότερη έρευνα και πορίσματα που θα ε, επηρεάζουν την κλήψη αποφάσεων. Ε, δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσαμε ή θα έπρεπε να αποφύγουμε μελέτες ε, που κάνει η βιομηχανία. Που μάλιστα η σοβαρή βιομηχανία, για να είμαι πολύ ομός, δεν έχει κανένα συμφέρον να φτιάχνει ψεύτικα αποτελέσματα. Μπορούν να υπερασπιστούν τα προϊόντα τους, αλλά δεν τους συμφέρει να έχουν πιο σοβαρά προβλήματα αργότερα με την ε, παροχή ψευδών στοιχείων. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια ισορροπία ανάμεσα στις δοκιμές και την, ε, της και την ε, δημοσίω χρηματοδοτούμενη έρευνα. Δεν θα σα εξηγήσω εδώ σε αυτή την αίθουσα τώρα υπερβολικά στοιχεία για το project του οποίου είμαι μέρος. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να συνδυάσει μοριακή επιστήμη και τοξικολογία ώστε να δώσει καινοτόμα μηχανισμούς και προσεγγίσεις ε, συγκεκριμένες. Εγώ υπερασπίζομαι αυτή την προσέγγιση, θα δούμε το αποτέλεσμα. Σίγουρα ε, απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο ηγείται το Πανεπιστήμιο του Λάιντεν και βέβαια δεν είναι μόνο για τους ενδοκρινικές διαταράχτες, αυτό είναι ένα κομμάτι μόνο. Αλλά δεν θα πω περισσότερα γιατί εγώ συμμετέχω σε αυτό το πρόγραμμα, άρα δεν είμαι αμερόληπτο. Θα αφήσω τον συνάδελφο τώρα να μας πει τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Ο καθηγητής Δίτριχ τώρα είναι θέμα οι ενδοκρινικοί διαταράκτε. <laughs> Okay, you put me on the, on, the spot then, okay. Βάλτε στον τοίχο τώρα. Δεν θέλω να απαντήσω έτσι με κατηγορηματικό τρόπο στον Αλμπέρτο. Δύο πράγματα. Είπατε αν διαφέρουμε ή αν νομίζω ότι διαφέρουμε και σε κάποιο βαθμό η κυρία Ροζιέρ το ίδιο ερώτημα έκανε. Επειδή παρουσιάσαν πολλά επιστημονικά στοιχεία, ίσως κάτι ξέφυγε από την προσοχή μας, ότι και οι τρεις ομιλητοί μίλησαν για ένα μείγμα για ένα συνδυασμό ε, ζητημάτων και ουσιαν και παράγοντων. Ο Αλμπέρτο, για παράδειγμα, είπε για αυτά τα λεγόμενα τα pathways, πόσο σημαντικά είναι τα μονοπάτια αυτά σε σχέση με την ποσότητα που ε, μπορεί να περάσει σε ένα έμβριο, για παράδειγμα. Ο Μάρτιν από τον Μπρουνέλ. Μίλησε πράγματι για αυτήν την, ε, αυτό το ιστρογόνο. Και ξέρουμε εκατομμύρια γυναίκες που έχουν ε, πάρει θεραπευτική αγωγή με διεθριστή λιβιστρόλη. 5% έχουν επηρεαστεί πιο πολύ, αλλά είναι... Μάλλον 5% είναι γυναίκες που δεν έχουν ε. To, to my colleague uh, uh or, um, member of Parliament, again, if we go back... Και το μεγαλύτερο ποσοστό δεν επηρεάστηκαν. Έγινε κάποια μελέτη πριν από κάποια χρόνια στις Πολιτείε. Mega Mouse Study, την είπαμε. Για να δούμε αν ε, το χλωρίχο νάτριο, το αλάτι, ε, συγγνώμη, αλλά να τα λέτε στο μικρόφωνο καλύτερα, αυτά που λέτε. Ναι, εντάξει. Απλά απευθυνόμουν στο κρατήριο στην αίθουσα. Λοιπόν, στη μελέτη αυτή για το τραπέζι αλάτι ε, βρέθηκε ότι είναι καρκινογόνο ουσία. Άρα θα έπρεπε να το απαγορεύσουμε. Αλλά η δόση είναι αυτή η οποία επηρεάζει. Ήταν ε, γελίο, γιατί δεν θα ξανακάναμε τέτοια μελέτη σήμερα. Γιατί το θέμα είναι η μελέτη, να μετράει τη σωστή δόση και βάσει τις δόσεις να κρίνει το κίνδυνος. Άρα δεν έχουμε και τόσο μεγάλη διαφορά. Έχουμε τις ε, ποσοτικές αυτές, ε, ε, την ποσοτική οδό, ε, quantitative adverse pathway, Μιλήσαμε για μείγματα, μιλήσαμε για φυσικές ορμόνες σε αντιδιαστολή με τεχνικά χημικά. Το θέμα είναι από πού και πάνω δεν είμαστε στα φυσικά όρια και από πού και πάνω υπάρχει κίνδυνος και πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσουμε από κοινού. Τα παιδιά μας, τα παιδιά μου είναι εκτεθειμένα σε καρκινογόνες ουσίες κάθε μέρα, σε αφλατοξόνες, σε αφλατοξίνες και παρόλα αυτά κοινωνικο-οικονομικά αποδεκτό υπάρχει κάποιο όριο. Μετά αρχίζει το πρόβλημα, αν υπερβούμε αυτά τα όρια που μας επιτρέπουν οι διατάξεις να αποσύρουμε από την αγορά τα προϊόντα που περιβαίνουν τα όρια. Κάποιος πρέπει να έχουμε εναρμόνιση, εγώ συμφωνώ αλλά για όλες τις ουσίες. Και να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος και ποια είναι η κατάσταση. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι εστιάζοντας σε πολύ λίγες ουσίες, χημικές ενώσεις, βλέπουμε μεν το δέντρο αλλά μας διαφεύγει το δάσος. Υπάρχει πληθώρα άλλων ενώσεων και ουσιών που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις και φυσικές ακόμα ο Αλμπέρτο που κάνει επιδημολογικέ μελέτε. Ναι, πράγματι μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν είμαστε πεπισμένοι ότι το πρόβλημα προέρχεται από τα συνθετικά χημικά. Εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα προέρχονται από φλεβονοειδή, από ζάχαρη και άλλα συστατικά ε, που παίρνουμε, επειδή άλλαξαν οι μας συνήθειες πολύ θερμιδική ε, μεγάλη θερμιδική πρόσληψη. Γι' αυτό και έχουμε και πολλούς ε, ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα παχυσαρκίας. Αυτά. Ευχαριστώ και ελπίζω να πάτε σε ερωτήσεις Είναι μαζί μας ε, online και η κυρία Μάρτιν. Υποθέτω ότι θέλετε κι εσείς να αντιδράσετε. Παρακαλώ όμως να μην μιλάτε γρήγορα. Συμφωνώ με τα άλλα μέλη του πάνελ. Συμφωνούμε δηλαδή ότι υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας και δεν υπάρχει μία ενιαία απάντηση για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα δημόσιας υγείας και δεν αφορά μόνο τις χημικές ουσίες. Επίσης, θα ήθελα να πω το εξής. Η χρονική στιγμή είναι πάντα πολύ σημαντική. Αν θυμάμαι, υπήρχαν ε, κάποιες αντιφάσεις για κάποιες εργασίες που έγιναν όσον αφορά ε, τους διαταράκτες για τις ε, εγγύους από την πρόσληψη κάποιων ουσιών όπως η διαθύστη βοστερόλη. Uh, Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν έχουμε πλήρεις και τέλειες γνώσεις για τις ιδιότητες ε, των ουσιών αυτών και τις ε, επιπτώσεις από την έκθεσή μας σε αυτές. Ως επιστήμονες, όντως ανακαλύπτουμε επιπτώσεις που δεν τις φανταζόμαστε και ε, απρόβλεπτες χημικές ουσίες εκεί που δεν τις περιμέναμε. Στην εφημερίδα εδώ το Σαββατοκύριακο, όπως ξέρετε, έγινε μεγάλη, δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα στην ύπαρξη ε, πλαστικών μικροϊλών στα μπουκάλια του εμφιαλωμένου νερού, τα πλαστικά. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθούμε την αρχή της, ε, for, της αλλά υπάρχουν ε, και άλλα κριτήρια, οικονομικά και πολιτικά, τα οποία οδηγούν αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Τώρα, η δημόσια έρευνα, η χρηματοδότησή της, νομίζω ότι είναι σημαντική. Δεν μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ. Και βεβαίως, εάν κάτι όπως η δημόσια έρευνα μπορεί να επηρεάσει την ε, έγκριση κανονισμών, την καλοδεχόμαστε. Θα πρέπει επίσης να δούμε ποια είναι τα συμφέροντα, τα ενδιαφέροντα, τις φαρμακοβιομηχανίες, όλων των εμπλεκόμενων τομέων και φορέων και οι επιπτώσεις των χημικών ουσιών στην ε, υγεία ξέρουμε ότι είναι πολλές. Θα πρέπει τα μηνύματα να αποστέλλονται σε όλους τους πολίτες μας ε, συνεχώς και να είμαστε πάντα προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει να αντιδράσει ο κύριος Ντίντριχ. Παρακαλώ σύντομα. Δεν θέλω να αντιδράσω σε αυτά που είπε συνάδελφο, αλλά μας ερωτήσετε τι γίνεται σε σχέση με την κανονιστική έρευνα και την επιστημονική έρευνα. Θα ήθελα να απαντήσω. Έχω την εντύπωση αυτή τη στιγμή ότι έχουμε επαρκή στοιχεία που μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε με την ε, ρυθμίσεις που πρέπει να έχουμε για, αυτούς, για αυτές τις ουσίες, για αυτά τα χημικά. Και ε, αν δεν έχουμε επαρκή στοιχεία πρέπει να δούμε πού έχουμε αβεβαιότητα για να επικεντρωθούμε και να προχωρήσουμε. Τώρα, όσον αφορά την ε, επιστημονική ακαδημαϊκή κοινότητα, ε, η έρευνα περισσότερο μας οδηγεί και δεν έχει να κάνει με το ρυθμιστικό σκέλος. Κάνουμε την έρευνα, δεν πρέπει να κάνουμε την έρευνα ως επιστήμονες. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να έχουν την εντύπωση ότι δεν έχουμε αρκετά επιστημονικά στοιχεία στη θέση μας για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Πιστεύω ότι έχουμε αρκετά επιστημονικά δεδομένα, όχι μόνο εδώ στην Ευρώπη, αλλά και στη ΣΥΠΑ. Διότι υπάρχει το ToxCast, το Read Across Program, όλα τα προγράμματα συνεργασίας τα οποία έχουμε, τα οποία είναι ευρύτατα τα διαδεδομένα, μπορούμε να συγκρίνουμε βάσεις δεδομένων, στοιχεία, έρευνες και είπε ο Ρομπέρτο ότι για ε, διάφορα ε, θέματα που αφορούν το θηροειδή και τη λειτουργία του Φερρυπίνα. Έχουμε στοιχεία επιστημονικά, αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε. Η επιστήμη είναι παρούσα με τα ευρήματά της, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να προχωρούμε. Ε, Ευχαριστώ. Έχουμε και τα Monsanto Papers όμως, που δεν μας καθησυχάζουν ότι δεν υπάρχουν και σφάλματα ε, στα ρυθμιστικά, στο ρυθμιστικό σκέλος. Ah, okay. <laughs> Uh, Bernard, you want to react from, from first panel? Θέλετε να απαντήσετε, ήσασταν στο πρώτο πάνελ, κύριε Bernard αλλά αν θέλετε, ναι. Σε πολλά θα ήθελα να αντιδράσω, αλλά τέλος πάντων. Θα εστιάσω σε ένα. Ο κύριος Ντίτριχ, μάλλον δεν καταλαβαίνει γιατί τη σφενόλη α θεωρείται άκρως ανησυχητική χημική ουσία. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Για να δείξουμε ότι μπορεί να υπάρχει συνένεση στην προκειμένη περίπτωση. Η Επιτροπή των Κρατών Μελών, μάλλον η Επιτροπή του Κράτους Μέλους, των κρατών μελών με πυρογνώμονες θα πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα για τη δυσφενόλη α. Όλοι συμφώνησαν, ομόφωνα πήρε, λήφθηκε απόφαση. Πηρεάζει αναπαραγωγικές ιδιότητες, μειώνει τη μνήμη, τις μασιακές δυνατότητες και μπορεί να βοηθήσει και σαν ανάπτυξη διαβήτη τύπου Β και άλλα ενδιαφέροντα Α. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Κύριος Μαντοβάνη. Ε, Αν μου επιτρέπετε να κάνω κόπι κόπ-πέ στον εαυτό μου. και να επανέλθω σε αυτό που είπε ο Ντάνιλ. Μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά, αλλά σε κάποια σημαντικά πράγματα συμφωνούμε. Ίσως ένα βασικό μήνυμα είναι να μην τα υπερπολι... τα πράγματα. Μπορούμε απλά να βελτιώσουμε. Σίγουρα έχουμε περιθώρια βελτιώσεων. Και να προστατεύσουμε το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. on, on scientific. Αυτό νομίζω ότι μπορώ να το πούμε, είναι ασφαλή από επιστημονική πλευρά. Δεν θα πρέπει να καθυστερούμε τη λήψη αποφάσεων και να περιμένουμε περαιτέρω έρευνα. Δυστυχώ, λέει ο πρόεδρο, δεν έχουμε ακόμη πολύ χρόνο, αλλά λίγο χρόνο έχουμε για το κρατήριο. Θα δώσω το λόγο σε τρει. Έναν βλέπω ήδη. Κάνα άλλο. Προσπαθώ απεγνωσμένα με τις ΜΚΟ να εργαστώ για τον τομέα αυτό. Το παράρτημα για τα κριτήρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και παραγνωρισμένο. Και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και ο ΕΚΑ ίσως θα έπρεπε να τα λάβουν αυτά υπόψη τους ότι το να λέμε ότι η βιομηχανία, τα αριθμιστικά, της τεστ, δεν θα αποβάλει σε συστημική ε, αξιολόγηση που είναι επιστημονική μέθοδος. Δεν είναι σωστό. Συστηματική αξιολόγηση σημαίνει ότι πρέπει να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, τα πάντα. Και αυτό δεν γίνεται. Thanks. Uh, professors, do you want to react? Θέλει κάποιος να απαντήσει. Is that, is that me you are addressing? Okay, thank you. Εμένα το λέγατε αυτό. Πρόεδρος. Οι άλλοι τα λένε μεταξύ τους. Εσείς, ε, εσείς που είστε μακριά, μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας. Ναι, σε ό,τι αφορά το σχόλιο για τη συστηματική αξιολόγηση, ναι, μπορώ κάτι να πω. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη ότι κατάλαβα βέβαια τι είπε ο κύριος. Μάλλον ήθελε να πει ότι δεν υπάρχουν ε, διαθέσιμα όλα τα στοιχεία. Κάποια δεν είναι διαθέσιμα ε, δημόσια. Και αυτό είναι ένα θέμα. Σε ό,τι αφορά τη βιβλιογραφία, το peer review, υπάρχει θέμα. Γιατί πράγματι πολλά δεδομένα δεν βγαίνουν ε, προς τα έξω. Και κάποια από αυτά που παράγει η ίδια βιομηχανία δεν διατίθενται. Δεν δημοσιοποιούνται. Από πλευράς διαφάνειας αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα μπορούσε όμως να προστατευτεί με κάποιο τρόπο η δημοτική ιδιοκτησία. Εφόσον αυτά τα δεδομένα πρέπει να δημοσιοποιηθούν γιατί έχουν επιπτώσει για τη δημόσια υγεία. Thank you so much. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Φτάνουμε στο τέλος αυτή της τόσο ενδιαφέρουσας και ουσιαστική συζήτηση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία τους όλους τους συμμετέχοντες, τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ε, αξιότιμους εμπειρογνώμονες και επιστήμονες για τις ε, πάρα πολύ πολύτιμες παρατηρήσεις για τη συμβολή τους και διότι σεβάστηκαν όλους τους κανόνες που είχαμε θέσει. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές που αφορούν το θέμα αυτό, δηλαδή το θέμα των ε, ενδοκρινικών ε, διαταρακτών και ε, ενός ασφαλούς περιβάλλοντος από χημικά. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και εστιάζουμε την προσοχή μας στον σημασία και στον ρόλο της έρευνας και της επιστημονικής εκτίμησης και αξιολόγησης για την προτροπή αυτών των κινδύνων από τα χημικά προϊόντα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους ε, επιστήμονες παρόντες, που είναι παρόντος. Είπατε ότι θα πρέπει να σας ακούσουμε, θα πρέπει να μας ακούσετε εσείς είστε όμως επιστήμονες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ μας, γιατί είμαστε πολιτικοί και εσείς έχετε ε, απόψεις που βασίζονται σε επιστημονική βάση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την συμμετοχή σας. Τώρα, το μήνυμα φαντάζομαι το έλαβε Επιτροπή. Και αυτό που ελέγχθη είναι ότι δεν ήταν και εξαιρετική η δική σας προσέγγιση. Θα ήθελα να πω ότι για διάρκεια αυτής της θητείας το 2016 συγκεκριμένα ε, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του όλου θέματος των ε, ενδοκρινικών ε, διαταρακτών. Ελπίζω ότι τέτοιου είδους προβλήματα δεν θα επαναληφθούν, διότι ακούσατε τι είπαν οι επιστήμονες, οι ειδικοί. Και βεβαίω, ξέχοντα τι επιστημονικέ γνώσει, πρέπει και εσεί να αντιδράσετε διαφορετικά και να ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα φτάσετε με μια τέτοια σχετική ε, ρύθμιση και έναν κανονισμό, θα έχετε την υποστήριξη και των δύο μεγάλων ε, πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε, σα ευχαριστούμε όλου για τη συμμετοχή σα.